να σας καλωσορίσω αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε το δεύτερο κομμάτι της συνεδρίασή μα. Ε, συνεδρίασής μας. Ε, έχουμε εδώ τον κύριο Πέκ από την ΙΠΙΚ. Ε, Ο κύριος Πέκ, εν πάση περιπτώσει, είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και θα πάρει μέρος στις ζητήσεις μας zusammenarbeit mit partnern jenseits unserer λοιπόν, η συγκήτρια έχει το λόγο, η κυρία Χέρτσοκ, για την στρατηγική προσέγγιση για έναν ασφαλή αηφόρο και ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό. Ε, ε, εν μέρει ακούσαμε τι είπε ο Πρόεδρος, γιατί αναβόσβηνα το μικρόφωνο του. έχουμε τελικώς την απόφαση και η έκθεση θα βασιστεί στον ε, κανόνα 15 με την ενισχυμένη ε, συνεργασία και την ε, καθήλυνα αρμόδια επιτροπή που είναι η Ήτρε. Αναγνώριση λοιπόν για το πιο σημαντικό μήνυμα που έχουμε σε σχέση με αυτό το φάκελο για την εξωτερική πολιτική ε, η οποία δεν είναι μεν πολιτική εξωτερικών υποθέσεων, αλλά είναι μια ε, διαδικασία για να έχουμε μια ενιαία αγορά στην ε, Ευρώπη, ενιαία αγορά και την ενέργεια. Έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν περισσότερη ασφάλεια σε σχέση με την ε, ενέργεια και την ε, ε, ασφάλεια παροχής στο μέλλον. Και έχουμε και το 194 που λέει ότι η ελληνική μπορεί να είναι καλύτερη έτσι, γιατί μοιραζόμαστε πολλά περισσότερα αντί να τα κρατάμε ο καθένας για τον εαυτό του. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας σας τι γνωρίζουμε από πλευράς χρονοδιαγράμματος. Ε, είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε όλοι. Έχουμε πρώτη η ανταλλαγή απόψεων σήμερα. Μετά θα συντάξω εγώ την έκθεση, η οποία θα στελεί ε, για μετάφραση μέχρι τον ε, Δεκέμβριο, οπότε θα έχετε, μέχρι τα Χριστούγεννα μάλλον, οπότε θα έχετε χριστουγεννιάτικο δωράκι στο δέντρο σας. Μετά 24-25 θα γίνει συνεδρίαση και θα συζητηθεί η έκθεση, 24-25 Γενάρη η ΑΦΕ, την ΤΕΒΕ και η ΙΝΤΑ επίσης περιμένουμε τις, να μας στείλουν τις ε, γνωμοδοτήσεις τους. Η γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ ε, είναι στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας. Οπότε όταν έρθουν οι τροπολογίες αυτής της Επιτροπής δεν θα ψηφίσουμε. Στις ε, τέλος Φεβρουαρίου μπορούμε να ψηφίσουμε την έκθεσή μας Μπορούμε να δούμε λοιπόν τις τροπολογίες και 21 μπορούμε να ψηφίσουμε την ε, ε, έκθεση. Ε, αν όλα πάνε καλά με τις μεταφράσεις και όλα αυτά, μπορούμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Θα σταματήσω εδώ, γιατί ήρθαμε σε επαφή με τους κοιόδης ηγητές και με τον Επιτροπό στην στο Στρασβούργο και θέλουμε να τονίσουμε ότι για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα έχουμε μία ακρόαση. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή πριν το τέλος του Γενάρη που είναι και η ε, προθεσμία για την αποβολή των ε, τροπολογιών, να γίνει αυτή η ακρόαση μαζί από κοινού και για την άλλη έκθεση που έχει κάνει ο συνάδελφος κ. Κάινς. Ε, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι καλό θα ήταν να ακούσουμε και τον Επίτροπο Έτινγκερ. Ο ίδιος είναι έτοιμος να έρθει, αν τον προσκαλέσουμε. Οπότε, Πρόεδρε, αν συμφωνήσετε και για την κρόαση, να στέλνουμε την πρόσκληση και στον ε, Δανό Υπουργό Ενέργειας, γιατί μάλλον όλο αυτό θα γίνει στα πλαίσια της ε, Δανέζικης Προεδρίας. Οπότε, να, τον, ε, να του στείλουμε την πρόσκληση. Επίσης, για το χρονοδιάγραμμα, καλό θα ήταν να γίνει αυτή η ακρόαση συμπεριλαμβανομένων και άλλων εμπλεκομένων φορέων. βεβαίως οι πρώτοι που θα ικανοποιηθούν φαντάζομαι αυτή την ακρόαση είναι οι ευρωβουλευτέ. Ε, παρακολουθούμε το τι γίνεται στο Συμβούλιο, στον τομέα αυτό και παρόλο που ε, τον Απρίλιο θα φτάσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση στην Ολομέλεια, φαίνεται ότι στο Συμβούλιο έχουν μια πολύ γρήγορη διαδικασία και το Συμβούλιο θέλει ήδη στις 24 του Νοέμβρη να ψηφίσει για το θέμα αυτό. Οπότε υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των δύο χρονοδιαγραμμάτων μας. Το Κοινοβούλιο βέβαια έχει την ε, δυνατότητα να ξέρει ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου για το θέμα αυτό και αν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Και επίσης αν υπάρχουν κοινά, κοινά, κοινές απόψεις, αν υπάρχει κοινό τόπος. Να ευχαριστήσω την κυρία Καρβάγιο, τον την κυρία Βαλεάν, τον κύριο Τόμσεν, που ήταν παρόντες στην πρώτη συνάντηση με τους α, ε, α, ε, ε, καθώς και τους άλλους δύο α, συναδέλφους που νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αν σας ενδιαφέρει μπορώ να σας πω και άλλα πράγματα αργότερα για το ποια είναι η θέση του Συμβουλίου, αλλά νομίζω ότι όλοι είχατε την ε, δυνατότητα να διαβάσετε το κείμενο. Το σημαντικό σε σχέση με την έκθεση αυτή είναι ότι πάνω από την ε, μισή ενέργεια που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται από τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι η, ε, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο. Οπότε είναι, είναι σημαντικό να έχουμε συντονισμό και να είμαστε συντονισμένοι σε, γενικώ σε αυτά που ξέρουμε για αυτές τις κυρίως διμερείς συμφωνίες ε, που ενισχύουν τις εισαγωγές μας. Νομίζω ότι είναι προτεραιότητα αυτή και θα ήθελα να πω ότι για την ε, γνωμοδότηση δική μας ε, η ιδέα ήταν ενός συναδέλφου βέβαια ε, θέλουμε να δούμε και τις τεχνολογίες της ενέργειας οι οποίες εξάγονται πάλι επί τη βάση διμερών συμφωνιών από την Ευρώπη προς άλλες χώρες, δηλαδή τρίτες χώρες. Και αυτό νομίζω ότι έχει αξία και θα πρέπει και ως προς αυτό να συντονιστούμε γιατί Αυτές οι ε, τεχνολογίες έγιναν με βάση την ε, έρευνα και τα εναντίστοιχη χρηματοδότηση που υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ώστε καλό θα ήταν να ξέρουμε κι εμείς τι ακριβώς εξάγουμε προς ε, τις τρίτες χώρες. Βέβαια το αν θα είναι πολιτική εξωτερική, εξωτερικών υποθέσεων ή ενέργειες ε, θα πρέπει να το συμφωνήσουμε, αλλά αυτή η εξωτερική διάσταση της ενέργειας πρέπει να αποτελέσει ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο ώστε να καταλήξουμε σε μια ενιαία αγορά ενέργειας και νομίζω ότι η έκθεσή μας πρέπει να το τονίσει αυτό. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εξωτερική πολιτική και την διάσταση αυτή ως τμήμα της πολιτικής εξωτερικών υποθέσεων. Ο δικός μας στόχος είναι να έχουμε μια ασφαλή παροχή ενέργειας για τον Ευρωπαίο πολίτη. Και βεβαίως όλα αυτά θα συνδυαστούν με άλλες ευρωπαϊκές ε, πολιτικές όπως το Connecting Europe Facility, ε, για η δίκτυα δηλαδή που θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από κάθε γωνιά της Ευρώπης και θα είναι διαθέσιμα στους πολίτες. Και βεβαίως η διασύνδεση όλων αυτών ε, θα, είναι, θα αποτελέσει ένα ακόμα πυλώνα της εκθεσής μας. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι διαβάζοντας την ανακοίνωση της Κομισιόν είδαμε ότι επικεντρώνεται κυρίως στην ε, πολιτική για, την, ε, για τις νότιες χώρες. Ε, νομίζω όμως ότι πρέπει να έχουμε λιγο, περισσότερο συνολική προσέγγιση γιατί το θέμα της ενέργειας είναι συνολικό, είναι παγκόσμιο ίσως, όχι μόνο περιφερειακό ή ευρωπαϊκό. Για παράδειγμα, το αέριο δεν έρχεται από, την, ε, από γειτονικές ε, χώρες, έρχεται από πολύ μακριά στην Ευρώπη. 16% της, ε, της χρήσης άνθρακα έρχεται από, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται από την Αφρική, ας πούμε. Οπότε όταν μιλάμε για το θέμα αυτό πρέπει να θεωρούμε και την Αφρική ως μια ήπειρο εταίρο. Πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα αυτό συνολικά από τον Βόρειο Πόλο μέχρι την Νότιο Αφρική και από την Ανατολική γειτονία μέχρι την, τις δυτικές υπήρους συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ της Νότιας Αμερικής και του Καναδά. Ε, ειδικά όταν μιλούμε για, για πόρους όπως ε, το αέριο, το φυσικό αέριο. Στον ε, Καναδά ας πούμε είναι σημαντικό αυτό και θα πρέπει ακριβώς να το δούμε ως ένα, ως ένα σύνολο. Αυτή λοιπόν είναι η α, ιδέα που θα ήθελα εγώ εδώ να παραθέσω κλείνοντας αυτή την έκθεση. Είπα και πάλι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τι γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται και με, και με τα εκτός και με τις εξαγωγές να μην επικεντρωθούμε μόνο στους ε, πόρους, τους ενεργειακούς, αλλά ε, να δούμε γενικώ και τις τεχνολογίες ενέργειας και η συνεργασία στον ε, τομέα της ενέργειας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ας πούμε, πρέπει να είναι ένα κομμάτι της προσέγγισής μας. Από τους πόρους που είναι η βάση μέχρι τους τελικούς χρήστες. Και πρέπει να δούμε και ποιος θα είναι υπεύθυνος γιατί. Στο παρελθόν θυμόμαστε όλοι ε, το αστείο που είχε γίνει για το ποιον θα πάρουμε τηλέφωνο όταν ε, υπάρχει θέμα με τα θέματα εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα ε, βλέπουμε ότι κινούμαστε προς την έβρεση ενός ομολόγου για τα θέματα ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιος θα είναι αυτό το άτομο, αν θα είναι δηλαδή ο εκπρόσωπο των εξωτερικών υποθέσεων ή ει ενέργεια. Εγώ σας είπα ότι αυτό νομίζω ότι εμπλέκεται στα χωράφια της ενέργειας και το Συμβουλίο προφανώς ενδιαφέρεται να ακουστούν και 27 φωνές ε, και νομίζω ότι ο δικός μας ε, στόχος θα πρέπει να είναι αν υπάρχουν 27 θέσεις με διαφορετικά εργαλεία, μάλλον θα πρέπει να έχουμε έναν που θα οργανώνει όλους αυτούς. Να μην ακούγεται δηλαδή σαν μια ορχήστρα που είναι ακούρδιστη και ο καθένας παίζει ό,τι θέλει, να υπάρχει ένας καλός συντονισμός από κάποιον, από έναν μαέστρο. Οπότε σημαντικό είναι να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε γιατί ακριβώς επειδή υπάρχει ε, ένδια πόρων, οικονομικών, ανθρωπίνων, ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε άμεσα ένα συγκεκριμένο δρόμο. Ε, δεν είμαστε εδώ για να τσακωθούμε, να βρούμε λύσεις προσπαθούμε και λύσεις λειτουργικές. Οπότε θα ήθελα να δω την άποψή σας, να μου πείτε και για το χρονοδιάγραμμα και για τα θέματα αυτά που πρέπει να συζητήσουμε. Και με θα ακούσουμε μεγάλο ενδιαφέρον και την Κομισιό και το Συμβούλιο. Αν εμεί ω μικρή ορχήστρα λοιπόν μπορέσουμε να κουρδίσουμε καλά τα όργανα μας για την ε, πολιτική και την ενέργεια, τότε ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε μάλλον θα είναι πιο ασφαλής, ώστε να επιτύχουμε το στόχο μας που είναι τελικά η ασφάλεια της ενέργειας για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτά. Από μένα ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε με τους ε, ομιλητές. Η κυρία Καρβάλιο πρώτα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πρέπει να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Χέρτσοκ, την εισηγήτρια, για τον τρόπο που συμπεριλαμβάνω όλα τα σημεία και κατά αυτόν τον τρόπο ξεκινά μια συζήτηση κατά αυτόν τον τρόπο των ενδιαφέροντα και είναι ανοιχτή αυτή σε όλες τις προτάσεις οι θα γίνουν στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιό καθότι κατά την άποψή μου η ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει είναι πλήρης νομίζω και καλά επεξεργασμένη Νομίζω πως πάει από, από τις πηγές ενεργείας που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης όλες οι γεωγραφικές επιτροπές, ε, περιοχές οικονομικές που υπάρχουν και όπως είπε η συγγήτρια πραγματικά ε, περισσότερο συγκεντρώνεται στις περιοχές εκείνες του Νότου. Επίσης δείχνουμε αυτή τη στιγμή την ασφάλεια, την ασφάλιση, την προμήθεια κλπ. Και όχι μόνο την εξασφάλιση προμήθειας αλλά όλους παράγοντες και αυτό είναι θετικό. Πρώτη σκέψη μου λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή θα είναι διμερής τα ισχυρά εκείνα σημεία τα οποία υπάρχουν και στο δεύτερο σημείο τις υποπεριοχές θα έλεγα, κύριες οι οποίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ότι είναι ε, συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση Κομισιό. Οι θετικές πτυχές τώρα είναι εκείνες οι οποίες δείχνουν κατά την άποψή μου ότι, ότι ενισχύει την συντονισμό της, της ε, πολιτικής της ΕΕ μεταξύ κρατών μελών και κομισιό στα πλαίσια των 27 χωρών. Νομίζω είναι κάτι αυτό πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και το γεγονός ότι η Ευρώπη θα είναι ικανή να μιλάει με μία φωνή θα δει σε εμά και σε όλη την Ευρώπη περισσότερη επίδραση που θα μπορεί να έχει και μία ισχυρή φωνή ε, σε όλο τον κόσμο. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης είναι και όπου μπορεί να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις είναι τα εξής. Πρώτον, η ανακοίνωση είναι πάρα πολύ λεπτομερής, γυτνιάζουν στις περιοχές, στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη βεβαίως, καθώς επίσης υπάρχει Λίγη αναφορά την Νότια Ατλαντικό, για παράδειγμα, όπως ελέγχθη προηγουμένως εδώ διαμέσου, την ενέργεια που έρχεται από την Νιγηρία, την Αγκόλα. Άρα οι χώρες του Νοτιού Ατλαντικού θα λέγαμε και του Ατλαντικού, Ατλαντικής θαλάσσης, δηλαδή της ωκεανού προφανώς. Ένα πράγμα το οποίο με εκπλήσει παρά η Νότια Αμερική, η οποία αποτελεί ένα μεγάλο χώρο, ευρύ χώρο, θα πρέπει να επιστηθεί περισσότερο η προσοχή μας και θα ήθελα αυτό να το υπογραμμίζω. Τρίτον, όσον αφορά τις ανερχόμενες οικονομίες, ε, Ινδία και Κίνα, κατά την άποψή μου θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στις ε, ανερχόμενες οικονομίες, ιδιαίτερα την Ινδία, και τις επιδρόσεις που θα έχει η Ινδία και πώς αυτό θα, θα το αντιμετωπίσουν στα επόμενα χρόνια. Υπάρχει ένα άλλο τελικά κεφάλαιο σε αναπτυσσόμενες χώρες, για τις αναπτυσσόμενες χώρες, νομίζω πως θα χρειαζόταν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την ανακεφαλαίωση και την συσσόρευση κεφαλαιοκή και πώς πραγματικά μπορεί αυτό να εξευρεθεί και πώς υπάρχουν υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες όπως στην Αφρική για παράδειγμα, πώς θα υπάρχει δυνατότητες για να υπάρξει εκεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και νομίζω πως η Ευρώπη πραγματικά μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο δεσμεύοντας αυτές τις χώρες για να υπάρξει μια καλύτερη. Ένα παράδειγμα μπορώ να σας δώσω που είναι η Μοζαμβίκη όσον αφορά το αέριο που ευρέθηκε. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομίζω πως πραγματικά υπάρχει όλο και περισσότερη επίδραση που έρχεται από την Νοτιοανατολική Ασία και νομίζω πως πραγματικά οι διασυνδέσεις που γίνονται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και πολύ περισσότερα παραδείγματα στην Αφρική, όπου πραγματικά εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ περισσότερο παρόντο και τη δυνατότητα να συμβάλλουμε και να έχουμε και πολύ καλές σχέσεις ε, με την Ιδία και τις χώρες εκείνες που ενδιαφέρουν αυτή την περιοχή. Επίσης, θα ήθελα περέντος να πω πως αυτές είναι οι πρώτες εντυπώσεις που ήθελα να καταθέσω εγώ ε, και σε σχέση με την ανακοίνωση της Κομισιόν. Θα ήθελα λοιπόν να συνεργαστώ στο μέλλον με την συγκίτρια και τους Σκιώδης και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Βάλιαν, σκιώδη συγκίτρια. Yes, uh, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να και μιλάω και πίνω, προσπαθώ να πάρω, να μου βάλουν τσάι μάλλον. Λαμπρά. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω μάλλον την κυρία Νομίζω πω θα είναι μια πάρα πολύ καλή εισηγήτρια. Θα έχει οργανώσει ειδικά ήδη, μα έχει βάλει στο κλίμα και εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονό ότι προσπαθεί όλου να μα βοηθήσει για να φτάσουμε σε ένα κοινό συμπέρασμα σε όλο το κοινοβούλιο βεβαίω και στην Επιτροπή μα, προτάσει οι οποίε έχουν γίνει και οι οποίε θα είναι η εποφελία όλων ημών και νομίζω πάει πέρα από ιδεολογίε, απόψει, θεωρίε και αφορά τη βιομηχανία. Ακόμη, ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω και το οποίο είναι σημείο κλειδί, το σημείο 1. Πράγματι, είμαι έτοιμη να δεχθώ τι προτάσεις Κομισιό με την προπόθεση εάν πείσει πω αυτά γίνονται για την αγορά. Διότι μέχρι στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε μια αγορά ενέργειας η οποία θα λειτουργεί σωστά. Κατά την δική μου άποψη λοιπόν οπτική γωνία νομίζω πως αυτό θα ήταν καλό αν γίνει για να εξασφαλιστούν υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας και φρονώ πως την ομόνια εγγύηση την οποία μπορούμε να έχουμε να βελτιώσουμε την αγορά. Βελτίωση της Πιστεύω πω αυτή είναι η οπτική γωνία από την οποία θα κοιτάξω εγώ αυτά τα αυτή την πρόταση που έχουμε να χείρασε. Βεβαίω υπάρχει κοινή, η, πολιτική, η κοινή πολιτική ενέργεια. Ε, δεν είχαμε μέχρι τούδε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν βέβαια λόγια που δεν είχαμε, αλλά νομίζω πως πραγματικά είναι ένα τομέα στον οποίο πραγματικά κράτη-μέλη είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους και δεν είμαι καθόλου πεπισμένη πως κάποιος είναι, κάποια αυτές τις χώρες είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τα προνοκτήματα τα οποία έχει για να αποδείξει την αγκή προς τις άλλες χώρες μέλη. Έτσι λοιπόν δεδομένο αυτό του σημείο θα πρέπει να παραδεχτώ ότι καταλαβαίνετε το τι λέω αυτή τη στιγμή και νομίζω πως έχουν τα πράγματα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να υπάρξει ένας το επί θέματος αυτού. Ένα άλλο σημείο το οποίο με ενδιαφέρει τα μάλα είναι το γεγονός ότι ενώ μιλάμε για την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν στη δικό μας μέσα στον κήπο μας. γιατί θα πρέπει να δούμε την εξωτερική διάσταση της χώρας. Ε, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι υποδομές και νομίζω πως η Κομισιόν, ξέρουμε αλλά η Κομισιόν ότι προτείνει υποδομές για την ενέργεια αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, διότι έτσι μόνο θα φτάσουμε στους στόχους στους οποίους έχουμε φτάσει. Αυτό από τη μία πλευρά. Από την άλλη μεριά θα οφείλω να ομολογήσω, εάν έτσι έχουν τα πράγματα των κρατών μελών σε σχέση ότι υπάρχουν ανάγκες για την ενεργειακή πολιτική, οι διαφορές είναι τόσο τεράστιες που θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας όταν αποφασίζουμε για ευρωπαϊκή πολιτική και για ευρωπαϊκό κανονισμό. Καθότι αυτό το οποίο φοβάμαι είναι, δεν πρέπει να αυτό το οποίο προσπαθήσω να ακολουθήσω και να αποφύγω να γίνει είναι ότι, ότι είναι θα πρέπει να θα δούμε τι θα δράσουμε εμείς ως παίκτες, ως πέσοντες στον τομέα στις ενέργειες. Διότι το ένα είναι πραγματικά να... Το ένα είναι πραγματικά να είμαστε παρόντες και να παίξουμε στη διακυβερνητική ως συμμετέχοντες και όχι ως παρατηρητές. Καφέ. Στο, στην αγορά της ενέργειας είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να ακολουθήσω και θα πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου. Αλλά νομίζω πως πραγματικά αυτό είναι ένα πρώιμο στάδιο της συζήτηση και βεβαίως θα υπάρξει η έκθεση και υπάρχουν εισηγητές οι οποίοι θα είναι πραγματικά των τεκτενωμένων και θα συνάδουμε αυτά. Ευελπιστώ λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχουμε το κείμενο να χείρα στο τελειωτικό και νομίζω πως τότε θα έχουμε την επόμενη φορά δηλαδή θα έχουμε μια, ένα ουσιώδη, ε, μια ουσιώδη ε, συζήτηση του θέματος. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε μέχρι τούδε. Αληθεύει πραγματικά ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να βρούμε μια συνένεση στην Επιτροπή μας. Αλλά το πιο σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει μια ισορροπημένη απόφαση μεταξύ οικονομικού μεταξύ της συμβα... Ε, συμβατικής ελευθερίας ε, της ασφάλειας, της των προμηθειών κλπ. Δεν δηλαδή είναι ισορροπημένο το κείμενο, να λαμβάνει όλους τους παράγοντες υπόψη. Για τα κράτη-μέλη, για όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω ε, πως είναι πολυμερές, πολυμερής η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Και πιστεύω πως το αέριο είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται των κανόνων της αγοράς. Και αφετέρου υπάρχουν ορισμένα μονοπόλια τα οποία χρειάζεται να υπαχθούν αυτά στο κοινοτικό δίκαιο. Συνεπώς πιστεύω πως δίνοντα τη δυνατότητα στην Κομισιόν τη δυνατότητα να δράσει είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν ισπανικά, λέει ένα ε, βουλευτή. Δεν ακούει τα ισπανικά, δυστυχώ. Υπάρχει πρόβλημα με τα ισπανικά, λέει ο πρόεδρο. Όχι, λένε οι Ισπανοί συνάδελφοι. Παρακαλώ, επαναλάβατε, κύριε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα μέχρι τούδε, ώστε να υπογραμμίσω ένα πράγμα. Λέω λοιπόν, υπάρχουν τα μυστικά του εμπορίου και τα δικαιώματα και τα προγράμματα που έχει η Κομισιόν να επιβάλλει να επιβάλλει έλεγχο από αυτό το θέμα. Αυτά λοιπόν, αυτή η ισορροπία μεταξύ των πρώτων και των δευτέρων που ανέφερα προηγουμένω, θα πρέπει να βρεθεί η ισορροπία, διότι διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα. Μερικά μονοπόλια θέλουν αυτή τη στιγμή να ξεφύγουν, να τι καπουλάρουν από αυτή την προσπάθεια των υπεθενικών Κομισιόν. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα πακέτο ενεργειακό εντό τη ΕΕ και το οποίο να υπάγεται σε όλους τους κανόνες οι οποίοι ισχύουν σε, αυτό, σε αυτή την αγορά που έχουμε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν εταίροι μας οι οποίοι είναι σοβαροί και οι οποίοι πραγματικά υπακούν σε αυτούς τους κανόνες στους οποίους έχει θέσει η Κομισιό. Καθώς επίσης ότι θα υπάρχει δυνατότητα αυτοί οι κανόνε να υπάρχουν και να είναι σοβαροί. Η έκθεση λοιπόν τη συγκέντρωση είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν καταστάσει τις οποίες είχαμε παλαιότερα στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη χώρα μου, διότι υπήρχαν κανόνες οι οποίες αναγκάστηκαν να τροποποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Κομισιό και νομίζω πως δεν θα πρέπει αυτό που συνέβη στη χώρα μας να συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Κύριε Καστίγιο, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφο καθώς και τους σκιώδεις εισηγητέ. γιατί πιστεύω ότι παρουσίασαν σήμερα κάτι πολύ καλό. Ανέφεραν τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μου θέματα μέχρι στιγμής. Επιτρέψτε μου όμως να, να δω τα πράγματα από μια πιο σφαιρική γωνία σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η πρόταση από την Επιτροπή πρέπει να ενταχθεί στην οπτική της ενιαίας αγοράς, ε, την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Η πρόταση για την εξωτερική διάσταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνδέεται με την οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς, όπως ανέφερε και η συγγήτρια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ουσιώδες ζήτημα. Υπό αυτήν την έννοια μπορούμε να δούμε την πρόταση αυτή ως ένα βήμα προς τα εμπρός προς ένα τρίτο πακέτο ενέργειας, προς ένα επόμενο πακέτο ενέργειας. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για την ε, μελλοντική ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Και αυτό θα μας οδηγήσει, αυτό μας φέρνει σε ένα τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, ε, δηλαδή κατά πόσο πρέπει ή δεν πρέπει να έχουμε μια ενιαία φωνή στην ε, Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας δρόμος, ένας δρόμος προς τον οποίο πρέπει να βαδίσουμε. Αλλά από την πλευρά του Κοινοβουλίου είναι σημαντικό να μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτό είναι ο στόχος. Προς αυτό το τέλος βαδίζουμε και υπό αυτή την έννοια πρέπει να εργαστούμε. Με αυτή την πρόπτικη πρέπει να ζητήσουμε συντονισμό για την οικοδόμηση μιας ενιαίας φωνής στο πλαίσιο αυτό. Ακόμα και αν σήμερα αυτό είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να το έχουμε στο νου. Δεν πρέπει να λησμονούμε τον ορίζοντα, γιατί αν δεν έχουμε ορίζοντα, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το στόχο, την ενιαία αγορά με ενιαία φωνή σε εξωτερικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να καλωσορίσω κάποιους ερευνητές εδώ στην, ε, στην Επιτροπή μας. Ε, οι οποίοι κάνουν μια ανταλλαγή, βρίσκονται σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής. Ε, καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στους κόλπους της ομάδας μας. Ευχαριστώ που μου το θυμήσατε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Βιντελ Κουάδρας έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ωραία είναι να αναγγέλλετε ότι υπάρχουν επισκέπτες. Γιατί άκουσα τόσο δυνατό χειροκρότημα και νόμιζα πως ήταν για μένα. Στην πραγματικότητα όμως είναι η συνάδελφος Χέρτζοκ είναι φαινόμενο. Τη συγχαίρουμε πριν καν δούμε την έκθεση. Πραγματικά, ε, είναι φανταστικό. Τρελό έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη στην κυρία Χέρτσοκ που ήδη τη συγχαίρουμε. Πραγματικά, είναι πολύ σπάνιο κάτι τέτοιο. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Είμαστε βέβαιοι ότι η έκθεση της θα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη σήμερα όμως μιλούμε για το κείμενο που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασφαλώς είμαστε ευχαριστημένοι που ήρθε αυτή η ανακοίνωση γιατί όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής. Ασφαλώς πρόκειται για θεμελιώδες ζήτημα, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί σήμερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει φυσικά να μιλούμε με ενιαία φωνή για να προασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας, ακόμα και στις ε, διμερής συνεργασίας. Πρέπει πολυμερείς συνεργασίες και συνομιλίες να αναπτύσσουμε, γιατί η ισχύς βρίσκεται εν τη ενώση. Ο καθένας μας μεμονωμένος είναι ευάλωτος, ενώ όλοι μαζί αποκτούμε δύναμη. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν, ας αποφεληθούμε από το γεγονός ότι μπορούμε να αποτελέσουμε μια δύναμη η ανακοίνωση την οποία λάβαμε με μεγάλη ικανοποίηση θα μας οδηγήσει πιστεύω σε μια αντικειμενική συζήτηση χωρίς ιδεολειψίες που θα δώσει καλύτερο, μεγαλύτερο περιεχόμενο στη διπλωματία μας στον τομέα της ενέργειας. Κάποιες παρατηρήσεις. Είναι σημαντικό για την ε, ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής της ενέργειας αλλά ακόμα πιο σημαντικό, γιατί είναι ε, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η συμπλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε να, έχουμε, να βρεθούμε σε θέση να διαπραγματευτούμε με τους εταίρους μας. Σίγουρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός τα τελευταία χρόνια με τα πακέτα, τα νομοθετικά για την ενέργεια Ωστόσο δεν μπορούμε ακόμη να μιλάμε πραγματικά για μια ενιαία αγορά ενέργειας. Για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο θα πρέπει να βελτιώσουμε τη δια... διασυνδεσιμότητα κατά τρόπο που να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι διακοπής του εφοδιασμού και όλοι μαζί να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στον κίνδυνο αυτό. Μια χώρα που αντιμετωπίζει τέτοιο κίνδυνο στον ανεφοδιασμό πρέπει να προστατευτεί. Πρέπει λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα. Επίσης, για την εγγύηση του ανεφοδιασμού, αυτό δεν το κάνουμε μόνο ε, κατασκευάζοντας ε, μεγάλες υποδομές όπως ο νότιος διάδρομος που φυσικά προσφέρει πλέον εκτήματα, δεν τα αρνούμε. Ωστόσο πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο εάν όλοι μαζί προάγουμε τις διαπραγματεύσεις, παρά ο καθένας μεμονωμένα. Πρέπει να συνεχίσουμε να πολλαπλασιάζουμε τους ε, του... τα... τα σημεία διανομής των ε, καυσίμων και πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι η ενέργεια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο. Ως εμπορικό όπλο και αυτό συζητήσιμο είναι. Πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν τον εσωτερικό συνδυασμό, συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και να καταφέρουμε να βρούμε το σωστό ενεργειακό μείγμα. Να έρθουμε σε επαφή και με τις τρίτες χώρες, σε πνεύμα αλληλεγγύης ασφαλώς, γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν συμφωνίες εποφελής για το ένα κράτος, αλλά ίσως επιβαρυντική για τα άλλα κράτη, πράγμα που δεν είναι αποδεκτό. Πρέπει να βρούμε επίσης ένα μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών για τις υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας. Τελευταίο σημείο που θα αναφέρω. Θέλω να στηρίξω, να, δηλώσω, να διαδηλώσω τη στήριξή μου σε αυτήν την ε, πρόταση της ε, Επιτροπής. Υπό την, ε, πιστεύω με κάποιες επιφυλάξεις ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας, θα διευρύνει το πλαίσιο αναφοράς, γιατί γίνεται πια αναφορά σε μια ανοιχτή αγορά. Και αν θέλουμε να έχουμε μια ασφαλή και βιώσιμη αγορά ενέργειας, χρειάζεται και μια νομοθετική σύγκληση. Είναι ευκταίο κάτι τέτοιο. Η ευρύτερη δυνατή νομοθετική σύγκληση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας ε, αυτοτελής σκοπός τον οποίο πρέπει να επιδιώξουμε και ολοκληρώνω. Όσο αφορά την εξωτερική πολιτική, δεν είναι πάντοτε εύκολο να βρεθεί κοινό στόχο μεταξύ των κρατών <coughs> μελών, γιατί οι γεωπολιτικοί παράγοντες της ενέργειας ε, παίζουν ρόλο. Υπάρχει αύξηση της ζήτησης και εξάντληση των καύσιμων πόρων για το μέλλον. Πρέπει να το έχουμε αυτό στο νου μας και πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Τώρα είμαστε σίγουροι ότι η έκθεση θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση γιατί αυτό μας ανέφερε και η ομιλήτρια. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είμαι ο μόνος που δεν έχει διαβάσει την έκθεση. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει καν ακόμα η έκθεση, οπότε μάλλον δεν την έχει διαβάσει και κανένας άλλος. Μια που έχω λοιπόν το λόγο να... πω και εγώ ότι στα καλύτερα χέρια έχουμε αφήσει την έκθεση αυτή, τη σύνταξή της, στα χέρια της κυρίας Χέρτσοκ. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε θα, και να, να είναι σίγουρη η κυρία Χέρτσοκ ότι θα την στηρίξουμε, θα τη στηρίξουμε η Ήτρε. όντως εδώ βρίσκεται σε ένα θέμα που είναι τη άμεση αρμοδιότητά τη. Εδώ μιλούμε για πολύ σημαντικές πολιτικές συνέπειες στον τομέα αυτό και για τώρα αν θα είναι η διάσταση εξωτερική της ενέργειας αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε από την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι οι χώρες ε, όπως η Σλοβακία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, ε, πάντα ήμασταν ε, πολύ ευαίσθητοι σε ό,τι αφορά την εξάρτηση από εισαγωγέ ενέργειας. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πάντα προκύπτει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και επίσης η διαφοροποίηση των εισαγωγών ενέργειας είναι εξίσου σημαντικό θέμα πάντα φοβόμαστε μήπως ε, η Ρωσία πάυσει, αναστείλει την παροχή αερίου. Είμαστε πραγματικά πολύ εξαρτημένοι από την χώρα αυτή και ελπίζω να υπάρξουν τα στοιχεία αυτά και στην έκθεση. Έχουμε και τον αγωγό Ναμπούκο. Ε, είναι σημαντικό για μας για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια, ένα βαθμό ανεξαρτησίας η ενέργεια μην χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό όπλο. Και επίσης ένα άλλο θέμα που, έχουμε, που έχω να θέσω. Ε, έχουμε και την πολιτική διάσταση της παροχής ενέργειας. Στον τομέα αυτό χρειάζεται να μιλάμε με μία φωνή. Είναι δύσκολο να, έχουμε, να το πράξουμε αυτό, γιατί ούτω ή άλλω η πολιτική ενέργεια είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμεί δεν έχουμε εδώ ενιαία ε, πολιτική ενεργειακή, οπότε πρέπει να συνεννοηθούμε. Ε, θέλουμε να επιτύχουμε μια εσωτερική αγορά, μια ενιαία αγορά ενέργεια, οπότε πρέπει να μιλούμε με μια φωνή. Και επίση πρέπει να πω ότι τον ε, τελευταίο καιρό έχουμε επεξεργαστεί πάρα πολλά έγγραφα για τον τομέα αυτό και καλό θα ήταν αυτή η έκθεση να περιλαμβάνει, να βασιστεί ίσως ε, σε αυτά τα έγγραφα. δεν έχει νόημα να δημιουργούμε μονίμως μια εξαιρετική μεν έκθεση, αλλά να κάνουμε σαν να μην έχει υπάρξει ξανά συζήτηση ποτέ για αυτό το θέμα. Ε, έχουμε και τα θέματα τα περιβαλλοντικά, την, ε, της αντιμετώπισης της, ε, των περιβαλλοντικών αλλαγών, την οικονομία του χαμηλού άνθρακα. Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, με όλα τα θέματα αυτά και νομίζω ότι θα πρέπει στην έκθεση να συμπεριληφθούν. Έχουμε καταλήξει και σε, πολλά, σε πολλές αντιφάσεις πολλές φορές. Έχουν γίνει έντονες συζητήσεις. Έχουμε συζητήσει για την πυρηνική ενέργεια. Ξέρω ότι είναι μικρό το βήμα που κάνουμε, αλλά πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα προς τα έξω. Μετά τη Φουκουσίμα, Βρισκόμαστε εδώ στην Ευρώπη σε, μεγάλη, σε πολύ δύσκολη θέση γιατί μιλούμε για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας πια και πρέπει να έχουμε μία ενιαία φωνή, πρέπει να κάνουμε κάτι με κάποιο τρόπο, δεν, πρέπει να, να μιλάμε καθαρά στο λαό. Το να μην μιλάμε ή να μιλάμε κρυφά μεταξύ μας δεν έχει νόημα. Εάν θέλουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον ε, με, εισαγωγούς, με εισαγωγικές εταιρείε ε, ή με εξαγωγικές εταιρείε, πρέπει να, συνεργαστούμε και στον τομέα της έρευνας για όλα αυτά. Αυτό δεν έχει βέβαια άμεση σχέση με την μεταφορά της ενέργειας, αλλά για να λυθούν τα προβλήματα της ε, παροχής ενέργειας, ε, νομίζω ότι ακριβώς και, ε, επειδή ο τομέας αυτός είναι σημαντικός, και η Ήτρα θα πρέπει να εμπλακεί για την μεταφορά, την ασφαλή της ενέργειας. Όλες αυτές είναι πτυχές ενός πολύ σημαντικού ζητήματος. Και ε, αν ε, μπορούσε να υπάρξει μια φράση μέσα σε αυτή την έκθεση που θα περιλαμβάνει αυτά τα θέματα, εμένα θα με έβρισκε σύμφωνο. Ευχαριστώ. Η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές καλές ιδέες. Πραγματικά ένα βήμα προς ε, μια πιο ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας. Υπάρχει ένα δίλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε καλές παραδοχές, έχουμε καλές θεωρίες, θέλουμε περισσότερη ολοκλήρωση, ενοποίηση, αλλά από την άλλη διακυβεύονται τα εθνικά συμφέροντα. Ε, καθώς θα προχωράει η σύνταξη της έκθεσης, ε, εγώ θα πρόσεχα όλος ιδιαιτέρως ορισμένα στοιχεία και κυρίως την υλοποίηση Έχω πολλές ανησυχίες ότι στο πλαίσιο των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο ε, πάντοτε αποδυναμώνονται στο τέλος οι ιδέες που υποστηρίζουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα πρέπει να, το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά. Να δούμε πώς θα υπερασπιστούμε καλύτερα τη θέση που αντανακλάει έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό να, να μοιραστούμε τις πληροφορίες για τις ε, διακυβερνητικές συμφωνίες. Αλλά υπάρχει και το θέμα της υλοποίησης. Έχουμε δει τι έχει συμβεί, τι συνέβη με το τρίτο πακέτο ενέργειας. Είδαμε πόσο ε, χρόνο διαρκούν οι διαδικασίες επί που εκκινούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πόσο δύσκολο είναι να συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη. Ε, είναι σημαντικό να επεκτείνουμε την κοινότητα της ενέργειας, την ενεργειακή κοινότητα. Αυτό είναι προς το συμφέρον των κυβερνήσεων. Η Επιτροπή έχει δίκιο όταν λέει ότι η ενέργεια θα πρέπει να είναι τμήμα της διαδικασίας ένταξης και συνεργασίας με τις υπόλοιπες χώρες επίσης κομμάτι των διαπραγματεύσεων ε, στον ΠΟΗ. Πολλά έχουν υποθεί για την ε, Ρωσία και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Υπάρχουν συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για το τρίτο πακέτο. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολες ε, οι διαπραγματεύσεις κατά καιρούς. Διαβάζουμε τα ανακοινοθέντα των Ρώσων ηγετών Κάποιο λέει ότι από αυτού λέει ότι δεν υπάρχει λόγος η Gazprom ή κάποια άλλη ρωσική εταιρεία να, να συμμορφωθούν με το τρίτο πακέτο, γιατί το πακέτο είναι ευρωπαϊκό. Το έγγραφο λοιπόν αυτό πιστεύω θα έχει ένα βάρος και πάνω στις συνεχιζόμενες αυτές διαπραγματεύσεις. Νομίζω πρέπει να υποστηρίξουμε να μην επιτραπούν παρεκκλήσεις, εξαιρέσεις από τις ρυθμίσεις για την εσωτερική αγορά. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι πραγματικά σημαντικό να αναπτύξουμε περαιτέρω τις ιδέες που περιέχει έκθεση και πρέπει να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην επιτρέψουμε την αποδυνάμωση των ιδεών αυτών και να σκεφτούμε και πώς θα τις υλοποιήσουμε, πώς να ενισχύσουμε την υλοποίηση αυτού του εγγράφου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πρώτες ύλες ε, μειώνονται συνέχεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πάρα πολύ σκληρά μέτρα έτσι ώστε να μπορέσει να εγγυηθεί την ανεξαρτησία της από την εισαγωγή ενέργειας. Είναι λοιπόν σημαντικό ό,τι υπάρχει στον τομέα αυτό να αποτελέσει τμήμα της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον και κυρίως στις διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών Επίση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τέτοια στοιχεία, ε, τέτοια δεδομένα, καθώ επίση και με συμφωνίε με άλλε περιφέρειες του κόσμου. Κάθε διμερή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτη χώρα ή άλλων περιφερειών του κόσμου πάντα θα πρέπει να, συμπεριλαμ... να ε, ορίζεται από το ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι ε, στον τομέα της ενέργειας και ότι αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να μπορούν να υποστηριχθούν από την ασκούμενη πολιτική. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Μήπως θέλει κάποιος από την Κομισιόν να παρέμβει. Σύντομα. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια καθώς και σήμερα το μέλλον που παρενέ, παρενέβησαν και τη θετική υποδοχή που έχουν κάνει στην ανακοίνωση Κομισιόν όσον αφορά την εξωτερική διάσταξη της πολιτικής ενέργειας. Ωραία, όπως υπογραμμήθηκε, που γραμμίστηκε. Η για πρώτη φορά αντιμετωπίσει συνολική προσέγγιση. Μια προσέγγιση θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και γι' αυτό προσπαθήσαμε να δείξουμε ποιε είναι οι προτεραιότητε όσον αφορά τη γυτνίαση καθώς επίσης και τις παραγωγικές χώρες, τις καταναλωτικές χώρες, τις ενερχόμενες χώρες μέσα σε αυτά τα πλαίσια της προσέγγισης θα πρέπει να δούμε προτεραιότητες καθώς επίσης να σκεφτούμε τη διαφορετική χρήση των οργαλείων τα οποία έχουμε να σε τεχνική υποστήριξη και διότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν σχέση με τη διαφορετική πτυχή που έχει ο κάθε εταίρος μας. Και θα θέλαμε από την άλλη μεριά να είμαστε πιο ισορροπημένοι. Βεβαίω υπάρχει ασφάλεια που θα πρέπει να γίνεται ω αφορά τους λογονάνθρακε. και αυτό είναι ένα θέμα που θα απασχολεί σε επόμενε δεκαετίε. αλλά θα πρέπει να θέσουμε και άλλα θέματα. Η επάρκεια, οι, ενέργειες, οι ανανεώμενες ενέργειες, το νομικό καθεστώς, αυτό όχι μόνο με τη στους χώρες και τους συμμάχους μας αλλά και τους εταίρους μας. Βεβαίω να δούμε τα θέματα που άπτονται με τα πυρηνικά ή την ε, εξόριξη offshore, στην ανοιχτή θάλασσα. Λοιπόν, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά συγκεκριμένα πράγματα και εδώ σε αυτό το συγκεκριμένα θέματα θα θέσω εγώ δύο θέματα κατά την άποψή μου, τα οποία τέθησαν και από τον εισηγητή γιατί είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο θέμα αφορά το συντονισμό. Ο συντονισμός στο πνεύμα της Κομισιόν δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί η δράση των κρατών μελών ή να, ή ο περιορισμός τους ή να περιοριστεί η δυνατότητα η δυνατότητα δράσεις των εταιριών της ΕΕ με τις, τις εταιρείες τρίτων κόσμων. Όχι, συντονισμό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια πληροφόρηση, μια ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών μελών και μεταξύ κυβερνήσεων. Πράγμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από μια ειδική επιτροπή και από τη δική επιτροπή για να δούμε πώς θα λειτουργήσει καλύτερα αυτή η εσωτερική αγορά της ενέργειας. Και δεύτερο σημείο που θέλω να πω, η συνέχιση αυτής της προσπάθειας μεταξύ όλων αυτών των προ... προθέσεων που έχουν τεθεί, καθώς επίσης αυτά τα οποία προβλέπονται από το 119 άρθρο της συνθήκης, δηλαδή να υπάρχει μία προοπτική της εσωτερικής αγοράς να λειτουργήσει σε αυτά και όλες οι προτάσεις οι οποίες γίνονται εδώ και οι δραστηριότητες να ακολουθούν αυτό το άρθρο. Χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί η συγγήτρια πραγματικά έδωσε αυτή την προοπτική και την ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και εσάς όλους. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κυρία Χέρτσοκ, θέλετε το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως πραγματικά κύριε βίδε Κάντα, συγγνώμη, αλλά νομίζω πραγματικά βρίσκομαι σε καλεστία, γιατί πήρα από τόσα καλά λαγιά. Αλλά όταν έγραψα την έκθεσή μου, δεν θα ήθελα να είμαι ούτε ελεφάντης ένα κροκόδιλος. Ο κροκόδιλος έχει μεγάλο στόμα και δεν έχει αυτιά. Και εγώ ήθελα να ακούσω πραγματικά αυτά τα οποία λέγονται εδώ πέρα. Και νομίζω πραγματικά η τελική θα πρέπει πέρα από αυτά που είπα να έχουμε μία φωνή και να ακουστεί αυτή μία φωνή προς τα έξω. Σαν κοινοβούλιο βέβαια σε αυτό. Γιατί ο ανώτατος χρόνος θα επιτευχθεί το 2040. Ο από τον Ντάρμιν είπε δεν είναι τούτε το ισχυρότερος, αλλά ο, ο ισχυρότερος και ο πιο έξυπνο, αυτό θα επιβεώσει είναι αυτό που θα αλλάξει μου λέει όπω το είπε αυτό, δηλαδή έτσι πιστεύω η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει και στο επίπεδο του πετρελαίου αλλά και τη νέα προσέγγιση που θα πρέπει να κάνει όσον αφορά την ενέργεια. Ο κ. Καρμπάγιο, ο κ. Μπάγια, ο κ. Σεντράκαν, ο κ. Κόνραντ και οι υπόλοιποι προλαλήσανες ο κ. Τουμασφόρο ο οποίο δεν ήταν εδώ αλλά Πιστεύω πως αυτό που είπε και ο Μισονός όσον αφορά την ασφάλεια για το πυρνικά εμείς πόσο μπορούμε να εξάγουμε το know-how, τη γνώση που έχουμε ε, προς τα έξω, αλλά παράλληλα αυξάνοντας την ασφάλεια που θα πρέπει να έχουν οι πυρνικοί μας αντιδραστήσεις εδώ στην Ευρώπη, νομίζω πως πραγματικά όλα αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα έγγραφο το οποίο θα τα συμπεριλαμβάνει και θα πάει προς την Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Εγώ παραμένω ανοιχτή αν θέλετε στις δικές σας προτάσεις. Έχετε όλοι εδώ ένα ρόλο να, παίξουμε, να παίξετε και όλοι μας έχουμε ρόλο να παίξουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την τελική σύνταξη αυτού του κειμένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ. «24 Ιανουαρίου» θα υποβληθεί η έκθεση και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Οπότε, κλείνουμε το σημείο αυτό της ημερής της διάταξης και πάμε στο σημείο 6. Επίσκεψη της Επιτρόπου, η οποία όμως θα έρθει και τέταρτο. Οπότε αν θέλετε να κάνουμε ένα σύντομο διαλυματάκι, αλλά αν θέλετε μείνετε κάπου εδώ κοντά, μην εξαφανιστείτε. Only a short break. Σύντομο διάλειμμα λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Το δεύτερο τμήμα του δεύτερου τμήματος της σημερινής συνεδρίασης. Να καλωσορίσουμε την Επίτροπο Κρούς, Επίτροπο για την ψηφιακή ατζέντα. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις πολλές φορές για το ένα ή το άλλο θέμα. Και πάλι έχουμε έτσι στα σπάργανα κάποια προγράμματα και χαίρομαι που είναι σήμερα εδώ η Επίτροπος Κρούς για να μας τα εξηγήσει, να τις θέσουμε ερωτήματα, να κάνουμε παρατηρήσεις. Παρακαλώ, Επίτροπε, έχετε το λόγο. Είναι μεγάλη μου χαρά, Πρόεδρε, να είμαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψα εδώ για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πολλές συναρπαστικές εξελίξεις. Υπήρξε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για την εξέλιξη της ψηφιακής κοινωνίας και την πρόοδο στην έρευνα κάτω από την τεχνολογία επικοινωνίας και πληροφοριών. Η Επιτροπή αυτή έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και βοήθησε με πολλούς τρόπους να δημιουργηθεί μια προηγμένη ψηφιακή κοινωνία στην Ευρώπη το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόσφατα κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για το πρόγραμμα πολιτικής για τις ραδιοσυχνότητες, το οποίο πρέπει να υιοθετηθεί τυπικά στις αρχές του επόμενου έτους. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την ενιαία αγορά για τις ε, ασύρματες ε, συσκευές, θα βελτιώσει τη διαχείριση του ευρωπαϊκού φάσματος και θα δημιουργήσει, θα διαθέσει μεγάλο χώρο των ραδιοσυχνοτήτων για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της τέταρτης γενιάς. Επίσης, θα αξιολογήσει τις ανάγκες ε, της μελλοντικές σε ραδιοσυχνότητες σε όλους τους τομείς και θα αυξήσει τη διαφάνεια στη διανομή ε, ραδιοσυχνοτήτων. Θα συνεχίσουμε ε, την προσήλωσή μας να υλοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερο τον κύριο Χόκμαρκ, τον εισηγητή και τον κύριο Ρεούλ, ο οποίος μαζί με πολλούς συναδέλφους από την Επιτροπή ξενύχτησαν πολλές μακρές βραδιές στη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου. Και αυτό με φέρνει σε ένα άλλο σημαντικό ε, πρόγραμμα, τον μελλοντικό κανονισμό για την περιαγωγή. Είμαι σίγουρη πως ε, σημερίζεστε την αποφασιστικότητά μου να επιφέρουμε σημαντικές, διαρκείς και δομικές αλλαγές στην αγορά για την περιαγωγή. Ξέρω ότι πρέπει να δώσετε στους ψηφοφόρους σας ένα απλό μήνυμα που να μπορούν να το ακούσουν. Οι χρήστες θέλουν πιο δίκαιες τιμές, πιο εύλογες ε, χρεώσεις και δεν θέλουν να φοβούνται ότι τα, ο τηλεφωνικός τους λογαριασμός στο εξωτερικό θα κοστίζει περισσότερο από τις διακοπές τους. Και εγώ το θέλω αυτό. Αλλά πρέπει να θεραπεύσουμε την νόσο, όχι απλώς να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα. Χρειαζόμαστε μια διαρκή λύση, η οποία να παρέχει ε, καινούριο και γνήσιο ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός έχει μειώσει τι τιμέ σε άλλες αγορές. Έχουμε τέτοια εμπειρία ε, στις αερομεταφορές για παράδειγμα, και σίγουρα θα μειώσει και τις τιμές της περιαγωγής. Θα απαιτηθούν για κάποιο χρόνο ανώτατα όρια τιμών, να μην ε, παρεξηγούμεθα, μέχρι να γίνουν αισθητά τα αποτελέσματα της ε, δομικής λύσης. Και σήμερα ε, εισάγουμε τέτοιες ανώτατες τιμές για την περιαγωγή των δεδομένων. Αλλά αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ορθό επίπεδο, να είναι ένα δίκτυο ασφάλειας για τον καταναλωτή, που αφήνει όμως περιθώριο για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Πολύ χαμηλά ανώτατα όρια δεν θα παράγουν σωστά αποτελέσματα και η εμπειρία μας έχει δείξει ότι δεν αποτελούν και την απάντηση. Για να επιτύχουμε ανοιχτέ αγορές και να υπάρχει πραγματική επιλογή για τον καταναλωτή, η ρύθμιση των τιμών δεν πρέπει να εμποδίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Εκτιμώ την ευρύτατη στήριξή σας για αυτήν την πρόταση. Ξέρω ότι έχουν εγερθεί κάποια ερωτήματα για την τεχνική υλοποίηση, για τα δομικά μέσα της, ε, τα δομικά μέτρα, τα διαρθρωτικά μέτρα της αποδέσμευσης. <clears throat> Έχουμε εξετάσει διαφορετικές λύσεις ε, υλοποίησης και είμαστε σε γόνιμες συζητήσεις με τον Μπέρεκ. Κάθε τεχνική λύση, συνδυασμός λύσεων, που οδηγεί σε εύκολες επιλογές για τους καταναλωτές και πραγματικό ανταγωνισμό είναι αποδεκτή για μας. Θα πρέπει να επιτύχουμε συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, γιατί αυτό θα εξασφαλίσει την υιοθέτηση πριν να εκπνεύσει ο σημερινός κανονισμός στο τέλος του επόμενου Ιουνίου. Και πραγματικά θα είμαι ευγνώμων αν μπορέσουμε όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Διαφορετικά θα υπάρξει ρυθμιστικό κενό. Ο καταναλωτής θα δει να εξαφανίζεται το δίκτυο ασφάλειας και θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο μέχρι να ριζωθεί ο ανταγωνισμός και η επιλογή. Και γι' αυτό, θα, ε, γι αυτό είμαι ευγνώμων για τη θετική σας στάση μέχρι στιγμής. Το άλλο σημαντικό ζήτημα πάνω στο οποίο δουλεύουμε μαζί είναι ο φορέας ενισά. Όπως ξέρετε, η φιλοδοξία μου είναι να ενισχύσω τον οργανισμό και να τον κάνω πιο αποτελεσματικό. Πρέπει να στηρίξουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα κράτη-μέλη και την κοινωνία γενικότερα, ε, για να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο διαδίκτυο, μεγαλύτερη από ό,τι σήμερα. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, η ΕΝΙΣΑ πρέπει να μπορεί να προσελκύει και να κρατήσει να διατηρεί στους κόλπους της τους ε, καλύτερους ειδικού για την ασφάλεια του ίντερνετ στην Ευρώπη. Δεύτερον, το προσωπικό και οι εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει να ε, έχουν άριστες συνθήκες για δικτύωση. Είναι ουσιώδες αυτό, ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να εκπληρώσει αποτελεσματικά την αποστολή του. Από την αρχή του Οκτωβρίου η ΕΝΙΣΑ έχει μια κινητή ομάδα βοήθειας με κέντρο την Αθήνα βοηθούν τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν την ικανότητά τους για ασφάλεια ε, του διαδικτύου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το κέντρο βρίσκεται στην Αθήνα. Και είναι ήδη αυτό μια θετική εξέλιξη. Και πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης νομοθετικής διαδικασίας είναι έτοιμο και διατεθειμένο να βρει λύσεις για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ελκυστικότητα του οργανισμού. Αυτό θα γίνει και μέσω διευθετήσεων ε, για, για να μπορέσουν οι επιχειρησιακές ε, υπηρεσίες να, παρέσ... παράσχονται σωστά από την Αθήνα. Είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε οποιαδήποτε βελτίωση ε, έρθει, από το, έρθει προς το μέρος μας πριν να υιοθετηθεί η κοινή θέση του Συμβουλίου. Η ασφάλεια του διαδικτύου, ωστόσο, δεν σταματά με πιο ισχυρή ενισά. Θα πρέπει... Είναι πολύ πτυχό το θέμα της ε, ασφάλειας. Εγώ προγραμματίζω μία φιλόδοξη στρατηγική πρωτοβουλία για την ασφάλεια του διαδικτύου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι το 2015 η στρατηγική μας, στρατηγική έχει θέσει ισχυρά οχυρωματικά έργα κατά των επιθέσεων και των διακοπών της λειτουργίας των δικτύων. Φυσικά, οι απειλές δεν έχουν σύνορα, γι' αυτό χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί με τρίτες χώρες για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν ασφαλή καταφύγια για αυτούς που επιτίθενται στο διαδίκτυο και για να προλάβει το να σχηματιστούν ειδικέ καταστάσεις σε κάθε χώρα, οι οποίες ε, γύρουν φραγμούς ε, για την βιομηχανία μας. Πρέπει επίσης να προστατέψουμε τους ευάλωτους χρήστες, να καταστήσουμε το διαδίκτυο πιο ασφαλές για τα παιδιά. Το να κάνουμε το διαδίκτυο έναν καλύτερο τόπο για τα παιδιά πραγματικά είναι μια προτεραιότητα της ψηφιακής, ε, του ψηφιακού θεμετολογίου. Το πρόγραμμα Πιο Ασφαλές Διαδίκτυο έχει δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα με κέντρα για το ασφαλέστερο διαδίκτυο για την ευαισθητοποίηση. Αλλά το ψηφιακό ε, περιβάλλον κινείται πολύ γρήγορα και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν και μπαίνουν στο διαδίκτυο ακόμη και από την ηλικία των 7 και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα κινητά τους και από τις κονσόλες των παιχνιδιών τους καθώς και από τους προσωπικούς υπολογιστές τους. Εν ώψη αυτών των αλλαγών, η Επιτροπή στους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική με σκοπό τα παιδιά να είναι ικανά να κάνουν τις, ε, την καλύτερη δυνατή και πιο ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Η στρατηγική αυτή θα έχει σαφείς στόχους και θα υλοποιηθεί μέσω ενός μείγματος πολιτικών, μεταξύ των οποίων μια ισχυρή συνιστόσα θα είναι η αυτορύθμιση. Για το σκοπό αυτό κάλεσα ένα συνασπισμό CEO από, την, από όλο τον κλάδο της τεχνολογίας ε, πληροφορικής και επικοινωνιών για να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε πολλούς τομείς, ε, μεταξύ των οποίων να αναφέρουν τις καταχρήσεις, να ενισχύσουν τον έλεγχο των γονέων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Το να γίνει το διαδίκτυο ένας πιο ασφαλής ε, τόπος απαιτείται για να έχουμε την εμπιστοσύνη των ε, χρηστών και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι εκ των ουκάνευ. Πιστεύουμε ότι μόνο μία πανευρω... ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για την ε, ηλεκτρονική ταυτοποίηση, αναγνώριση και υπογραφή θα φέρει την απαραίτητη συνοχή για τις ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και θα τονώσει και την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό στο δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους θα παρουσιάσω νομικά μέτρα ε, για να μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν μια ηλεκτρονική ταυτότητα για να έχουν πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες και μια πρόταση για να αναθεωρήσουμε την ε, οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή. Η επαναχρησιμοποίηση κρατικών δεδομένων, δημόσιων δεδομένων προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη. Η αξία της αγοράς για την επαναχρησιμοποίηση δημόσιων δεδομένων υπολογίζεται στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά τα έμεσα ωφέλη μπορεί να φτάνουν και τα 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ωφέλη των ανοιχτών δεδομένων δεν είναι μόνο οικονομικά. Ε, μπορεί αυτό να βοηθήσει τους πολίτες να συμμετέχουν στην κοινωνία και την πολιτική ζωή, να αυξήσει την λογοδοσία και την διαφάνεια, να βελτιώσει την αποτελεσματική και τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής. Και γι' αυτό προτείνουμε μια φιλόδοξη και συνεκτική Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ανεχτών Δεδομένων. Θα προτείνω τροπολογίες για την ε, οδηγία, για την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και για την επικαιροποίηση των κανόνων για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2012 θα ξεκινήσει η πύλη ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα καταστήσει τα δικά μας δεδομένα προσβάσιμα και χρησιμοποιήσιμα. Ο τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών επίσης ε, έχει και... είναι και πράσινος τομέας. Ε, μπορεί να βελτιώσει την αποδοτική χρήση της ενέργειας, να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και να έχουμε αποταμιεύσεις ε, ύψους του 15%. Η πρωτοβουλία αποδοτική χρήση της ενέργειας είναι η κύρια συμβολή της πολιτικής της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών για την τήρηση των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα. Για το σκοπό αυτό ε, και το πρόγραμμα συχνότητας εξετάζει τη δυνατότητα διάθεσης φάσματος για έξυπνα ενεργειακά δίκτυα και έξυπνα συστήματα μέτρησης. Ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε μια δημόσια διαβούλευση στο τέλος του έτους. Ανάλογα με τη δημόσια διαβούλευση και την ε, αξιολόγηση επιπτώσεων θα αποφασίσω τι θα κάνουμε στο τέλος του 2012. Ε, θεμελιώδες για μας είναι να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και την απροτεία μας στη βιομηχανία και για μας πολύ σημαντικό είναι η έρευνα που βρίσκεται από πίσω η πρότασή μας για τον προϋπολογισμό μετά το 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντανακλά τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο μέλλον της Ευρώπης μέσω της στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας. Η νέα προσέγγιση της ολοκληρωμένης έρευνας και καινοτομία με ορίζοντα το 2020 χέρι ευρεία υποστήριξη από τι εμπλεκόμενε πλευρέ, όπω έχει δειχθεί από την ανταπόκριση στην πράσινη βίβλο. Ο ορίζοντα 2020 έχει τρει στόχου. Πρώτον, την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Δεύτερον, ε, βιομηχανικά πρωτεία και ανταγωνιστικό πλαίσιο. Τρίτον, αριστεία με, επί τη βάση της επιστήμης. Είναι τρεις στόχοι ψηλού επίπεδου που αμοιβαία ενισχύουν ένα τον άλλον. Για να μεγιστοποιήσουμε την επίπτωσή τους, θα, συμμετέ, θα συνδυάσουμε την χρηματοδότηση του ορίζοντα 2020 με άλλες πηγές. Για παράδειγμα, τα περιφερειακά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, ε, τη χρηματοδότηση από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από την πλευρά μας, τονίζουμε τη σημασία της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών ως μια τεχνολογία που επιτρέπει πολλά πράγματα, ξεκλειδώνει και ανοίγει το δρόμο για πρόοδο και σε άλλους τομέας. Ταυτόχρονα θέλουμε να απλοποιήσουμε την πρόσβαση, να μειώσουμε το διοικητικό βάρος, να προσελκύσουμε τους καλύτερους ερευνητές και τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις. Θέλουμε να έχουμε ενιαίο σύνολο κανόνων για τη συμμετοχή και απλο, απλούστερους κανόνες χρηματοδότησης. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια απλή αρχιτεκτονική προγράμματος. Το ορίζοντας 2020 ε, είναι επίσης ταγμένο στην ενίσχυση της χρήσης των ΣΔΙΤ στα κράτη-μέλη. Αυτό θα απαιτήσει βέβαια ισχυρότερες δέσμευση από τα κράτη-μέλη όσο αφορά τις οικονομικές τους δεσμεύσεις και την ευθυγράμμιση των ε, εθνικών διαδικασιών. Φυσικά δεν αγνοούμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ε, η οικονομική κατάσταση για την Ευρώπη είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει, ότι δεν οφείλουμε να δράσουμε. Αντίθετα, πρέπει να οικοδομήσουμε ένα εύρωστο πλαίσιο πέρα από την ε, τρέχουσα οικονομική ε, αδυναμία. Και για μένα υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Ο τομέας ε, της τεχνολογίας των πληροφοριών, ένας από τους λίγους που πραγματικά μας δίνει ανάπτυξη που πολύ τη χρειαζόμαστε. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε νέα τόνωση στην ανάπτυξη. Γι' αυτό θα ήθελα να σας μιλήσω για μια νέα και πολύ συναρπαστική νομοθετική πρόταση, την το επωνομαζόμενο Connecting Europe Facility, ένα εργαλείο για τη σύνθεση της Ευρώπης. Ο στόχος μας κάθε Ευρωπαίος να γίνει ψηφιακός είναι κλειδί για την ικανότητα της Ευρώπης για καινοτομία και ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει την παροχή πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας και προσβάσιμη ε, οικονομικά υποδομή, όπου και αν είναι κανείς, όποιες και αν είναι οι ικανότητές του, όποια και αν είναι τα μέσα του. Οι παράγοντες αυτοί είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, τη στήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Για να το κάνουμε αυτό, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει πολύ στη νέα υποδομή για το γρήγορο ίντερνετ. Πέρα όμως από τους παραδοσιακούς παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, το Connecting Europe Facility συνενώνει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πιθανών επενδυτών, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις κοινή ωφέλεια, θεσμικοί επενδυτές, κατασκευαστές εξοπλισμού και κρατικές αρχές, σε συνδυασμό με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, το μέσο αυτό θα αυξήσει τις πιθανότητές μας να επιτύχουμε τους στόχους του 2020 για το γρήγορο ίντερνετ. Τώρα, για το μέσο αυτό, το Connecting Europe Facility. Το ψηφιακό κομμάτι έχει δύο στόχους. Πρώτον, να υποστηρίξει την εκδίπλωση ευρυζωνικού υψηλής συχνότητας. Δεύτερον, <clears throat> να παρέχει ζωντανά, σε ζωντανή σύνδεση με το ίντερνετ, δημόσιες και δικτυωμένες υπηρεσίες. Συνήθως οι υπηρεσίες αυτές σταματούν στα σύνορα. Εμείς θέλουμε να είναι προσβάσιμες σε όλους που διαβιούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε να επενδύσουμε 9 δισεκατομμύρια ευρώ από τους πόρους της Ένωσης σε αυτές τις ζωτικής σημασίας ψηφιακές υποδομές. Αναμένουμε ότι τουλάχιστον 9,2 για την ακρίβεια δισεκατομμύρια. 7 από το μέσο, τα οποία θα μοχλευθούν μέσω των νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων για τη στήριξη επενδύσεων άνω των 50 δισεκατομμυρίων και έως 100 δισεκατομμυρίων ε, ευρώ σε ευρυζωνικές υποδομές υψηλής συχνότητας. Αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό όταν μιλάμε για τέτοια χρηματικά ποσά. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 45 εκατομμύρια νοικοκυριά ή πάνω από 100 εκατομμύρια πολίτες και καταναλωτές οι οποίοι συνδέονται θα μπορέσουν να συνδεθούν σε ευρυζωνικά συστήματα υψηλής συχνότητας χάρη στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υπόλοιπα χρήματα θα στηρίξουν τις υποδομές, τις ευρωπαϊκές δημόσιες και δικτυωμένες ε, υποδομές υπηρεσιών. Καταλαβαίνω ότι αποτελεί πρόκληση να πείσουμε τα κράτη-μέλη και τις τοπικές αρχές να ξοδέψουν χρήματα για την τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών. Δεν είμαι τυφλή στι πολλέ ε, συγκρουόμενε προτεραιότητες που έχουν. Ωστόσο, σε μια κατά τα άλλα βραδιπορούσα οικονομία, η τεχνολογία αυτή μας υπόσχεται καλές αποδόσεις για τις επενδύσεις μας και τα ωφέλη τα οποία μπορούν να μοχλευθούν από το βασικό κεφάλαιο στις υποδομές είναι δεκαπλάσια. Γι' αυτό σας καλώ να διαδώσετε αυτό το θετικό μήνυμα πίσω στις χώρες σας και να βοηθήσετε να βάλουμε την Ευρώπη πίσω στο δρόμο προς την ανάκαμψη. Να μην ε, έχουμε μόνο μια ζωφερή άποψη για το μέλλον, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, προβλέπουμε να κάνουμε τον απολογισμό για το ψηφιακό θεματολόγιο μέσω ενός ευρύτατου διαλόγου με τις εμπλεκόμενες πλευρές. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας να κινηθούμε προς την ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα συνεχίσουμε να, αντιμετω... να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε τομεί όπου οι αποσπασματικές εθνικές πολιτικές απαιτούν συντονισμένη ευρωπαϊκή ανταπόκριση και να αξιολογήσουμε τι συμπληρωματικέ δράσεις μπορούμε να είναι όριμες για περαιτέρω δράση. Η ψηφιακή συνέλευση 2012 επίση θα, δώσει, θα βάλει το λιθαράκι της σε αυτή τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Χαίρομαι γιατί άκουσα ότι η Επιτροπή Ήτρε συμφώνησε να στη... μας στηρίξει στη διοργάνωση αυτή τη ε, ψηφιακή συγκέντρωση εδώ στο Κοινοβούλιο. Και έρχομαι στο τέλο. Μπορείτε ε, ίσως ε, για την επόμενη ψηφιακή συνέβρεση να συγκεντρώσετε κάποια επιτυχη... επιτυχημένα ψηφιακά παραδείγματα με βάση το τι συμβαίνει στις εκλογικές σας περιφέρειες. Θα ήθελα πραγματικά να έχουμε κάποια παραδείγματα βιτρίνας να δείξουμε για να εμπνεύσουμε. Ε, έτσι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια πιο στενή σχέση με τους ε, πολίτες, τους Ευρωπαίους, τους ψηφοφόρους σας, τους εκλογείς σας και να αναδείξουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για την βελτίωση της καθημερινότητάς μας μέσω της ψηφιακής ατζέντα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω εξ όλων την Επίτροπο για τις ε, Πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσε, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις πριν ξεκινήσουμε τη γενική συζήτηση. Καταρχάς για την περιαγωγή. Είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση και όλοι οι συναδελφοί ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για αυτές τις νέες τεχνολογίες ε, και τη χρήση τους το συντομότερο δυνατόν. Γιατί εκεί έχουμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω ότι και για το ΕΝΙΣΑ θα υπάρξει μεγάλη υποστήριξη. Γι' αυτό καμιά φορά είναι δύσκολες συζητήσεις, γιατί ε, δεν σκεφτόμαστε μόνο πρακτικά, ε, αλλά πώς μπορούμε να έχουμε και τα δίκτυα και τους και τους ε, εμπειρογνώμονες και πολλές φορές αυτές οι συζητήσεις είναι και φορτισμένες συναισθηματικά. Γι' αυτό πρέπει όντως να δούμε τον πυρήνα εδώ του θέματος και να δείξουμε την απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε ε, άνθρωποι που έχουν ε, υψηλέ προδιαγραφές να μπορούν να εργαστούν σε τέτοιες θέσεις. Ξέρω ότι είναι σημαντικό για εσά, ξέρω εξίσου πόσο δύσκολο είναι. Η κυρία Καστίγιο παίρνει πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο που είναι παρούσα σήμερα και μας παρουσιάζει την πρόταση της ε, Κομισιόν για το πρόγραμμα του 2012 και όλα όσα έχουν να κάνουν με την Ευρώπη του 2020. Ε, έκανε μια πολύ καλή ανάλυση της κατάστασης και μας έδειξε και τις προοπτικές που υπάρχουν Νομίζω ότι επικεντρωθήκατε περισσότερο στα, στην πιο σημαντική πτυχή του θέματος. Το πώς δηλαδή μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, που στο τέλος είναι αυτό που έχουμε περισσότερη ανάγκη και αυτό που θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε τις ε, τεχνολογίες ε, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών. Αν δείτε τι έχει γίνει φέτος το 2011 και τα όσα έχει προτείνει η Κομισιόν και τα έχουμε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο, το γεγονός ότι εξευρέθη συμφωνία με το Συμβούλιο ε, είναι πολύ θετικό. Έχουμε το πακέτο για τα, για τα δίκτυα και παρό, παρά τις αρχικές ε, δυσκολίες που υπήρξαν, τα, το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό στη συμπεράσματα του Συμβουλίου. Όπως ε, έχετε πει κι εσείς, Έχουμε και το θέμα της ασφάλειας σε σχέση με τον ΕΝΙΣΑ. Έχουμε και την πρόταση για την περιαγωγή που συνδέεται άμεσα με τους καταναλωτές. Οπότε νομίζω ότι γενικώ η εικόνα είναι αρκετά θετική, αρκετά αισιόδοξη. Τώρα θα μπούμε στο 2012 και είναι ακόμη πιο επίγον ε, για όλους μας να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια σωστή δομή για, την, ε, για τις τεχνολογίες πληροφορικής και τις τηλεπικοινωνίες. Και επίσης ε, πρέπει να δούμε την ε, νέα γενιά των ε, τηλεπικοινωνιών και με, με, εξέπληξε το γεγονός ότι μια πτυχή του προγράμματος αυτού λείπει. Το cloud computing, το οποίο ε, ανακοίνωσε η Κομισιόν και είπε ότι το 2012 θα υπάρξει μία πρόταση, προς το τέλος μάλλον του 2012 είπε η Κομισιόν. Μάλλον είναι αργά για να υποβληθεί μια τέτοια έκθεση τότε. Και όχι μόνο είναι αργά, αλλά δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται και στο πρόγραμμα καν του 2012. Γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασία. Νομίζω ότι έχει ε, καταδειχθεί σαφώς ότι η χρήση του cloud computing έχει τεράστιες επιπτώσεις σε αυτούς τους τομείς. Ε, η Κομισιόν λέει ότι η ΕΠΑ υπέβαλαν ήδη τη δική τους ε, ομοσπονδιακή ε, στρατηγική για το cloud computing τον Φλεβάρη. η οποία μάλιστα θα εφαρμοστεί και άμεσα, μέσω του cloud computing. Οπότε, γιατί η δική μας η αντίστοιχη στρατηγική λύπη, χρειάζεται ένα πλαίσιο στρατηγικής ε, αντίστοιχο. Και τελικά τι θα γίνει, θα καταλήξουμε σε κάποια νομοθεσία. Χρειάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του cloud computing στην ε, Ευρώπη. Οπότε αυτό είναι αυτό που με ανησυχεί εμένα περισσότερο. Τα υπόλοιπα τα είπατε πάρα πολύ σωστά και οι εξηγήσει σας επίσης ε, είναι πολύ σαφείς και πιστικές, αλλά αν δεν έχουμε αυτό το πυλώνα, ε, τότε νομίζω ότι ε, είναι λίγο ετοιμόρροπο το όλο οικοδόμημα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, η συνάδελφος Χολ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο πράγματα ήθελα να τότσω. Αυτές οι υπηρεσίες όσον αφορά το περιοχή για το ε, ψηφιακό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει και πραγματικά πιστεύω ξέρω ότι αυτοί θέλετε να καταργήσετε αυτές τις διασυνοριακές αλλαγές Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που έχουν γίνει αυτή τη αναφορά το θέμα αυτό καθώς απερινώ τις ηλεκτρονικές υπογραφές διασυνδέοντας τις διάφορες στρατηγικές που υπάρχουν, στρατηγικές για τα παιδιά κλπ. Πολλά πράγματα που υπάρχουν κατά πόσο. Η Κομισιόν προτείνει άραγε ότι μπορούμε να έρθουμε αυτή τη στιγμή με ένα δρομολόγιο, θα ένα χάρτη όπου θα υπάρθουν 100% πλήρωση και να συμπεριλάβει ένα είδος ομπρέλας που θα συμπεριλάβει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή επιτάπητος και το οποίο μπορούν να συμπεριληφθούν αυτά επόμενους μήνες. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία μέσω δορυφόρου, αυτές οι προτάσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων Ο σκοπός είναι να γίνει πολύ πιο γρήγορα, υπάρχει ταχύτητα πιο γρήγορα σε αυτά και μπορεί να βοηθεί στα κράτη-μέλη να είναι πιο συντονισμένα. Διαρωτώ με λοιπόν κατά πόσο, μπορείτε να πείτε και για αυτό το θέμα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτής της απόφαση του Συμβουλίου κατά πόσο θα είναι δυνατότητα να οθήσουμε να πάει πολύ γρήγορα ή υπάρχει ακόμη πραγματικά πολλή δρόμος και ότι θα είμαστε καθυστερημένοι όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Τέλος. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές διαδόσεις ψήθυροι για αυτό το θέμα και διαρωτώ με κατά πόσο είδατε, αισθανθήκατε τις συνέπειες που υπάρχουν αυτού του την άδεια που θα πρέπει να έχει τις άδειες που θα πρέπει να έχουν αυτές οι, οι κινητές τηλεφωνίες μέσω δορυφόρου και θα μπορούν να τα πουλήσουν αυτά τα δικαιώματα τα δορυφορικά σε μια τρίτη χώρα. Εάν αυτό συμβεί, ποια θα είναι το αποτέλεσμα όσον αφορά την απόφαση που θα έχει λεφθεί για την εφαρμογή τους στην Ευρώπη, εφόσον πουληθούν βεβαίω σε τρίτες χώρες και πώς αυτό πραγματικά θα έχει μία επίπτωση και βεβαίως ένα, μια επιπτωση και βεβαίω ενα επί των πολιτών της ΕΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μέρκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε για την παρουσίαση ε, που κάνετε όσον αφορά το προγραμματίο το 2012. Καταρχήν θα ήθελα να σα πω τα εξή ότι η αγορά, η ψηφιακή αγορά, η κοινωτική ψηφιακή αγορά δεν λειτουργεί καλά. Όσον αφορά την περιαγωγή, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να γίνει μια νυχτή όλα αυτά. Βεβαίως, διαρωτώ με κατά πόσο θα έχουμε ένα μια κοινή αγορά όσον αφορά την περιαγωγή. Σκοπός σας είναι, αλλά πραγματικά πιστεύετε ότι μπορούμε... Δεν πρέπει να πηγαίνουμε αργά-αργά, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μία απόφαση η οποία θα εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες. γιατί και πότε θα έχουμε αυτή την ψηφιακή αγορά η οποία θα είναι ενιαία μεταξύ των iPhone ή άλλων κινητών δεν γνωρίζω και δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή εγώ να κατεβάσω μουσική γιατί ξέρετε υπάρχουν δικαιώματα προστασίας των συνθετών και ξέρω ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κοινή ε, πολιτική. Υπάρχουν διαφορετικές προεπτικές από χώρα σε χώρα αλλά και τι θα κάνετε σε αυτό το θέμα και τι θα κάνετε ακόμη πώς θα κάνει το διαδίκτυο το ίντερνετ δηλαδή πιο ασφαλές για τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας καίει ειλικρινά, αλλά πώς, πώς θα το κάνετε. Είπατε ότι τα παιδιά των 7 ετών είναι ήδη στο διαδίκτυο αυτό είναι χαρούμενο αφενός, αλλά αφετέρου είναι και ανησυχητικό, διότι θα πρέπει οπωσδήποτε να, να παρακολουθηθούν αυτά τα παιδιά όταν πηγαίνουν πραγματικά πάρα πολύ νωρί στο ίντερνετ. Και μια ειδική ερώτηση, η οποία άπτεται το ευρωπαϊκό partnership όσον αφορά τον εταιρισμό ε, που ξεκινήσατε εσείς με το συναδελφό σας της Κομισιόν. Ξέρετε αυτό ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο αν δεν κάνω λάθος, άμα δεν απατώμε και και ακούσαμε πολύ λίγα πράγματα να λέγονται για αυτό το θέμα. Κατά πόσο διαρωτώμε υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι απτά. Τι θα κάνετε και τι πραγματικά θα λανσάρετε για το 12 όσον αφορά το θέμα αυτό. Τέλος, η, η, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η e-government, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι μια, μια ιδέα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν ξέρω πραγματικά εσεί τι σκέψει να κάνετε συγκεκριμένα. Ο επόμενος παρακολουθεί, παρακαλώ, Τσίκερσον. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Χαίρετε κύριε Επίτροπε και είμαι χαίρο, που είστε εδώ. Θα μπορούσα άραγε να δείξω δύο θέματα. Το, πρόξο, το πρώτο είναι το ενίσα. Ασπάζουμε τα αισθήματα που εκφράσατε, τι απόψει όσον αφορά αυτή την οργάνωση. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη οργάνωση καθώς επίση και οι όρια εργασία για το προσωπικό. Υπάρχουν πραγματικά δύο αντιδράσεις όσον αφορά αυτό το θέμα. Ξέρετε, οι λεπτομέρειες πάντα βρίσκονται, ο διάβολο βρίσκεται στις λεπτομέρειε. και οι συζητήσει συνεχίζονται όσον αφορά τις πτυχές τη εντολής που έχει και την εντολή η οποία έχει, ιδιαίτερα έγινε μια συζήτηση όσον αφορά την έκταση, τη χρονική έκταση αυτή της εντολής και συζήτηση όσον αφορά τη θέση, το χώρο, τον τόπο αυτής της της εταιρείας αυτής του πρακτορείου πού ακριβώς θα εγκατασταθεί. Ξέρετε, έχουμε ανεπίσημες συζητήσεις με τις ελληνικέ αρχές πριν δύο εβδομάδες περίπου. Ωστόσο, για λόγους δεδομένων των συνθήκων πριν δύο εβδομάδες για την Ελλάδα ήταν... Ε, δεν είναι εκπληκτικό ότι δεν καταλήξαμε αλλά ωστόσο υπάρχει δυνατότητα να επανέλθουμε στο θέμα αυτό πριν είναι πολύ αργά. Αν κοιτάξουμε πραγματικά τα διάφορες τροπολογίες οι οποίες έχουν καταθέσει συνάδελφοι όσον αφορά τους, κατα... τους στόχους, τον κατάλογο και τους σκοπούς αυτής θα πρέπει να τους να τους σταθεροποιήσουμε, να τους συγκεντρώσουμε, να τους οθήσουμε κατά τέτοιο τρόπο για να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Βεβαίως υπάρχουν λόγοι για τους οποίους πραγματικά αναβάλαμε για να υπάρχει ένα Το χρονοδιάγραμμα μας δίνει ευτυχώ αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε και να επανέλθουμε σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία κρεμούν και εγώ το αναφέρω αυτό στην έκθεση και νομίζω πως στο τέλος θα φτάσουμε σε μια άριστη, καλύτερη, βέλτιστη απόφαση. Εν πάση περιπτώσει το Γιάννιο και νομίζω ότι μετά τις διακοπές του τέλους του χρόνου θα είμαστε καλύτερη θέση και φόρμα για να αποφασίσουμε. Πώς έχει αυτή, αυτή ήταν μια ενημέρωση όσον αφορά για το Ρώμη τώρα. Θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζουμε την η άποψη ότι θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός όσον αφορά την περιαγωγή, την εγχώρια περιαγωγή και την εξωτερική, γιατί πραγματικά περνάμε σε πολύ τεχνικές, τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά την περιεγωγή στο επίπεδο της βιομηχανίας σε σχέση πώς μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός και πώς μπορεί να επιτευχθεί. Και είναι ένα θέμα πολύ καυτό, αλλά είναι σημαντικό γιατί χρειαζόμαστε να βρούμε τρόπο να βάλουν περισσότερο ανταγωνισμό στην αγορά, όχι πλήρη. Και έχοντας υπόψη ε, ότι η παλαιότερη νομοθεσία προσπάθησε να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά τα κατάφερε. Βεβαίως, φτάσαμε σε ένα σημείο γιατί πραγματικά υπήρχε προηγουμένως ένα σοκ που, σοκ που δημιουργείται λόγω της πληρωμής που γινόταν ε. Βεβαίως θέσαμε ένα όριο πλαφόν όσον αφορά το θέμα για σε λιγότερο κόστος που κοστίζει σήμερα, ωστόσο είναι ένας στόχος αυτός που σας αναφέρω για τη μείωση δηλαδή, τον οποίο τον ασπαζόμαστε όλοι ευελπιστώ. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να γίνει αυτό ο διαχωρισμό και νομίζω πως πραγματικά ότι θα είναι ένας επικοδομητικός τρόπος για να προχωρήσουμε και σε αυτό το τομέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μανουέλ παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που η παρουσίασή σας ήταν πάρα πολύ σημαντική και τις παρατήρησεις οποίες έχετε και μπορώ ήδη να σας πω ότι σε μεγάλη πλειοψηφία Αποδεχόμαστε αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως. Ωστόσο, ορισμένε ερωτήσεις που θέλω να σα θέσω για θέματα τα οποία θα εξεταστούν εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα οποία ενδεχομένω δεν έχουν τεθεί και αναπτυχθεί ικανοποιητικά, επαρκώ. Για το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα ψήφισμα που έχει σε σκοπό σε ένα σε μια ουδέτερη θέση καθώς επίσης και ενός πακέτου που έχει σχέση με τις τηλεπικοινωνίες συγγνώμη, καθώς επίσης και ένα ψήφισμα στο οποίο αναφέρονται οι ανησυχίες που έχουμε σε σχέση με πρακτικές οι οποίες μπορούν να αναπτύσσονται και οι οποίες εμποδίζουν την πρόσβαση σε ορισμένε υπηρεσίες. Και ε, έχουμε πει ότι το δίκτυο θα πρέπει να είναι ουδέτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις προτάσεις οι οποίες κάνατε για την βελτίωση. Και η ερώτηση που θέλω να θέσω είναι η εξή συγκεκριμένη. Η Κομισιόν κατά πόσο έχει σκοπό αυτή τη στιγμή να παρέμβει θα πάρει μέτρα νομοθετικά άλλα τα οποία μπορούν να τη βοηθήσουν. Διότι αυτά είναι στα, στα χέρια των κρατών μελών, γιατί και στα κράτη μέλη μπορεί να υπάρχουν πλαίσια νομοθετικά διαφορετικά από χώρα σε χώρα, πράγματα τα οποία θα είναι ενάντια σε αυτή την ενιαία προσπάθεια που γίνεται για την ψηφιακή. Ερχόμαστε όσον αναφορά το ΕΝΙΣΑ, το Κοινοβούλιο. Ξέρετε, σήμερα έχουμε μία γνωμοτότηση που υιοθετήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Επίσης, μία άλλη η οποία θα γίνει στην Επιτροπή Ελευθεριών καθώς επίσης και τις νομοθετικές εκείνες ε, διατάξεις οι οποίες οι οποίες αντιτίθεται σε οποιαδήποτε πειρατεία. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε την ε, εγκληματικότητα στο διαδίκτυο. Όλα αυτά τα μέτρα δεν συνδέονται μεταξύ του. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα καλύπτει όλες αυτές τις προσπάθειες για να κάνει το ίντερνετ, το διαδίκτυο πολύ πιο ασφαλές. Εμείς ε, ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών προτείναμε να υπάρχει ένας συντονιστής όσον αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο, για να υπάρξει ένας συντονισμός, για να υπάρχουν οι δραστηριότητε, οι πρωτοβουλίες οι οποίες γίνονται εκ μέρους των διαφορετικών φορέων και σωμάτων για αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω την άποψή σας γι' αυτό όσον αφορά τη δημιουργία ενός τέτοιου συντονιστή ο οποίος θα συμπεριλάβει όλες αυτές τις προσπάθειες που, γίνεται, που γίνονται και πού θα βρεθεί αυτή η προσωπικότητα που θα αναλάβει αυτή την εκπόνηση και πού θα μπορούσε να είναι σε ποιο τομέα θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί. Επίσης είμαι πάρα πολύ σύμφωνος, σύμφωνη με αυτό το οποίο είπατε και αυτό που είπε ο πρόεδρο. Θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Και όσον αφορά το πρόγραμμα του, με ορίζοντο 20, 2020, Πάντα εκτιμούσα εγώ ότι η ισότητα των δυνατοτήτων θα πρέπει να είναι ένας από τους πυλώνες για την υλοποίηση της αγοράς, της ψηφιακής αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο που πρέπει να είναι αποτελεσματικό, ευέλικτο. Και κάνετε μία παρουσίαση των διαφορετικών τομέων και αυτό ήταν πολύ σαφές. Μία ακόμη ερώτηση στο αυτό θέμα. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνίας θα παίξουν ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό στο 2020. Αλλά θα ήθελα να σας το εξή ερώτημα. Κατά την άποψή σας, το 20 πώς πραγματικά μπορεί να μειώσει τις διαφορές που υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή από χώρα σε χώρα. Κατά πόσο αυτό θα επιτευχθεί μέχρι το 20. Κύριε Νταλιάν, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Εκτιμώ πολύ ότι ξεκινήσατε την διαβούλευση για τις μεθοδολογίες για την κοστολόγηση και τις τιμές για την πρόσβαση και την μη διακριτική μεταχείριση σε αυτή την πρόσβαση. Το εκτιμώ γιατί θεωρώ ότι είναι έτσι, θαραλέο βήμα για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό για το ψηφιακό θεματολόγιο τώρα για το 2012 και το σχετικό πρόγραμμα εργασίας. Εκεί δεν αναφέρεται η συνέχεια, η παρακολούθηση αυτών των δημοσίων διαβουλεύσεων, ούτε αναφέρεται καμία ημερομηνία που να προβλέπεται για την δημοσίευση των ε, υπερχόμενων συστάσεων. Γιατί ακριβώς δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Ε, οι συστάσεις για το θέμα αυτό νομίζω ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το, η, τα διευρυζωτικά δίκτυα προσφέρονται σε ε, σωστές τιμές ε, και να εξασφαλίσουμε την ε, πρόσβαση των, των, στις επόμενες γενιές δικτύων. Επίσης, η Κομισιόν θα αναλάβει συγκεκριμένη δράση στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας για να βελτιώσει την ενιαία αγορά για τις των, των τηλεπικοινωνιών και τις επιχειρήσεις, γιατί νομίζω ότι και αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγικότητα ε, σε μια περίοδο που προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε την ε, ανάπτυξη στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για την περιαγωγή που πρότεινε η Κομισιόν. Είχα την ευκαιρία ήδη να σας πω ότι όντως πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη διαρθρωμένη λύση, γιατί εμείς έτσι καταλαβαίνουμε τον κανονισμό ότι είναι μια διαρθρωμένη λύση. Είναι μια διαρθρωμένη λύση. Μπορεί να μην είναι αυτή που θα προτιμούσαμε όλοι, αλλά είναι μια λύση. Ερώτημα όμω. Γιατί αν αποσυνδέσουμε τι υπηρεσίε περιαγωγή τις διατηρούμε ουσιαστικά συνδεδεμένες σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή γιατί ο πελάτης δεν μπορεί από την υπηρεσία περιαγωγής ή μάλλον γιατί αυτό δεν είναι κομμάτι της λύσης σας να αγοράσει μια υπηρεσία περιαγωγής σε ένα διαφορετικό κράτος μέλος από τον παροχό που έχει στο εθνικό του κράτος μέλος γιατί εγώ έτσι καταλαβαίνω τον όρο Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Μπορείτε να μου πείτε γιατί αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στη λύση που προτείνετε. Για τα υπόλοιπα ξέρετε ότι πάντα υποστηρίζουμε την Κομισιόν για θέματα ICT γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μέσο. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρβάλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο που έκανε τόσο λεπτομερή περιγραφή του προγράμματος Εργασία για το 2012. Εγώ θα επικοινωθώ στον ορίζοντα 2020. Χαίρομαι που τονίσατε το θέμα της ε, απλούστευσης της αρχιτεκτονικής των απλών κανόνων, απλής δέσμης κανόνων και αναφέρατε και την ανάγκη για παραπληρωματικότητα, για συμπληρωματικότητα και συνέργειες με, την, με τα διαρθρωτικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό συνάδει απόλυτα με αυτό που συζητούμε και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Να σας ε, ρωτήσω κάτι για τις προτεραιότητες όχι για τον ορίζοντα 2020, αλλά αναφέρατε στην ομιλία σας το, τις τεχνολογίες ICT και τον τομέα τη ενέργειας, τα εφή δίκτυα, τους εφή μετρητέ κτλ. Είναι ένας τομέας αυτός πολύ ευρύς και πολύ σημαντικός για την Ευρώπη, για τις μεταφορές. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα για τις προτεραιότητες που βλέπετε στα, στα πλαίσια των ε, προτεραιοτήτων για το, 2020, για το 2020. Ε, στο πρόγραμμα πλαίσιο, ο τομέας των ICT έχει συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία αφορούν τις μελλοντικέ αναδυόμενες τεχνολογίες και οι οποίες μπορούν να δώσουν πολύ καλά αποτελέσματα. Όπως είπε και η συνάδελφος Φιώνα, ε, ακούγεται έτσι εδώ ότι το πρόγραμμα αυτό θα ε, ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Υπάρχει μια θετική πτυχή το ότι θα διευρυνθεί έτσι σε όλους τους τομείς της επιστήμης και αυτό είναι καλό. Αλλά το κακό είναι ότι σπάει ο δεσμός με, τον, με την όλη εφαρμογή. Η ιδέα αυτή βεβαίως είναι πολύ σημαντική για την εφαρμογή του ICT, οπότε εσείς πώς βλέπετε αυτό τον σύνδεσμο που υπάρχει με την έρευνα από κάτω προς τα πάνω θα συνεχίσει να υπάρχει με την όλη εφαρμογή. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόγια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ την Επίτροπο και έχω έντονο ενδιαφέρον για όλες τις προτάσεις που μας παρουσίασε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας πάνω σε δύο στιγμή και θα ζητήσω και μια ενημέρωση. Καταρχήν υπάρχει το, ένα κεφάλαιο στο ψηφιακό θεματολόγιο το οποίο αφορά την απέτηση ορισμού μιας νέας κατηγορίας, ενός νέου σώματος δικαιωμάτων, να τα ονομάσουμε έτσι η προστασία του καταναλωστή ε, θέλουμε να είναι μέρος όλων αυτών των ρυθμίσεων για το ψηφιακό θεματολόγιο και τις τηλεπικοινωνίες. Ε, μερικές φορές γίνεται λόγος για καταναλωτή, άλλες φορές για παιδιά, άλλες φορές για το πρόσωπο, για τον πολίτη, αλλά ίσως αυτή η πρωτοβουλία <clears throat> την οποία μας αναφέρατε, πώς θα ορίσει τα δικαιώματα των πολιτών στην ψηφιακή εποχή. Ε, αναφέρατε το ΣΕΦ το Connecting Europe Facility. Και μεγάλο μέρος της σημερινή μας συνεδρίασης ε, αφιερώθηκε ακριβώς στη συζήτηση αυτού του μεγάλου προγράμματος το οποίο είναι πολύ φιλόδοξο από μία άποψη. Από μια άλλη άποψη, μοιάζει να μην είναι τόσο σαφές ως προς την αποτελεσματικότητα των μέσων και των ε, χρηματοοικονομικών μέσων που χρησιμοποιεί χρηματοδοτικών μέσων. Αυτή η στόχη που δώσατε και δώσατε και αριθμούς για το πόσα άτομα, πόσες ε, οικογένειες θα έχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες και θα συνδεθούν με αυτές θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, ε, γιατί είστε και γνώστης του θέματος όλοι μιλούν για αυτό το ε, αποτέλεσμα μόχλευσης, το, το πολλαπλασιαστικό. Ε, δεν ξέρω, συνήθως ε, δεν έχουμε και μεγάλη εμπιστοσύνη στις, ε, στους ε, δημόσιους υπαλλήλους όταν πενεύουν τα εργαλεία τους. Θέλουμε να δούμε και θα με ευχαριστούσε πάρα πολύ εάν μας λέγατε πώς ακριβώς συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αυτό το εργαλείο το οποίο αναφέρατε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να έχετε υπόψη και την ώρα. Ε, στις ε, και μισή θα διακόψουμε. Θα είμαι σύντομος. Ακούστηκε το θέμα της εσωτερικής αγοράς ε, και ένας ε, μεγάλος όμιλος κατασκευής ε, κινητών τηλεφώνων και τάμπλετς λέει ότι δεν, έχει την, δεν παρέχει την σχετική υπηρεσία όταν μπει κανείς στην ιστοσελίδα του και αυτή, καμιά φορά αυτή την εντύπωση έχω και εγώ στην Ευρώπη ότι δηλαδή δεν είναι κάτι διαθέσιμο αν ας πούμε πάει κανείς να αγοράσει μουσική ή αν θέλει να στείλει μουσική διασυνοριακά, δεν μπορεί να το κάνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί έχουμε ε, τους ε, κανόνες της εσωτερικής αγοράς και σίγουρα, κυρία Κρούς, ξέρω ότι εσείς είσαστε η σωστή, ώστε, η σωστή επίτροπος για να ικανοποιήσετε αυτό το αίτημα. Έχουμε μια, ένα ψήφισμα επίσης για την ουδετερότητα των δικτύων και είπαμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί η ανάπτυξη Κάποιοι τομεί τομείς της των παλιών βιομηχανιών είναι, έχουν αποδυναμωθεί πλέον και τώρα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία αν το διαχειριστούμε το θέμα καλά. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει η ίδια διαχείριση και να υπάρξει ουδετερότητα των δικτύων παρόλο που μπορεί να δημιουργείται εντύπωση ότι πλήττεται η ουδετερότητα των των δικτύων. Ε, αν και στην ε, Ολλανδία οι νομοθέτες το έχουν λύσει το πρόβλημα αυτό ό,τι αφορά τα κινητά. Έχετε σκεφτεί, έχετε αναλάβει κάποια δράση ώστε αυτό να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ε, χώρες Είπατε για την ευρωπαϊκή στρατηγική, για την, για την ασφάλεια του ίντερνετ. Αυτό είναι σημαντικό οι πελάτες δεν πρέπει να έχουν φόβο να μπουν στο δίκτυο και να ψωνίσουν, να κάνουν αγορές ε, διασυνοριακά, αλλά καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι στην Κομισιόν ε, έτσι δημιουργούμε φόβο σε κάποιες ε, συζητήσεις και ερχόμαστε έτσι με διάθεση τιμωρίας και κάποια πράγματα πρέπει να παραμείνουν ε, εγκρυπτό. Ε, δεν θα πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό. Ε, την, ε, τη δύναμη που έχετε τη χρησιμοποιείτε με τον σωστό τρόπο γιατί μερικές φορές υπάρχουν κανόνες εκεί που δεν χρειάζεται και απλώς προκαλείται φόβος για τους καταναλωτές και έτσι δεν νομίζω να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη από τους καταναλωτές ώστε να δημιουργήσουμε και την ψηφιακή, τους ψηφιακούς πολίτες. Οπότε ξαναρωτώ και πάλι για την ψηφιακή ιστορική αγορά που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να υπάρχει σε όλα τα κρατημέλη και για την ε, ουδετερότητα των δικτύων για να ενισχύσουμε την ε, ανάπτυξη και να δώσουμε τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν καινοτόμα προϊόντα και να μπορούν να τα παράσουν μέσω διαδικτύου. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, συνάδελφοι, έχουμε συντονιστές. Και επίση η, συνάδελφ, η, η Επίτροπος πρέπει να απαντήσει κιόλα. Και έχω και άλλους που ζητούν το λόγο. Η κυρία Χέρτσοκ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, Πρόεδρε. Όλα τα νομοθετικά θέματα έχουν τεθεί. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι για το, για το ρόλο των γυναικών στους Financial Times του Σαββατοκυριακού υπήρχε ένα άρθρο για τις ε, πέντε γυναίκες ε, ηγετικές μορφές, ε, πολύ λίγες από την Ευρώπη, ελάχιστες στην ψηφιακή εποχή. Συνήθω αυτέ οι τεχνολογίε αφοσιώνονται στου ε, άντρε. Νομίζω ότι πρέπει να σπάσουμε αυτό το κατεστημένο και η, ε, η Κομισιόν είχε μια πολύ καλή πρωτοβουλία με τι γυναίκε στην ε, ψηφιακή εποχή, στο ICT. Αν δείτε και πόσε γυναίκε είμαστε εδώ μέσα στην αίθουσα. Νομίζω ότι καιρό είναι πια να ασχοληθούμε και με αυτό. Το Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει, αλλά πρέπει να μα πείτε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε. Ε, ο συνάδελφος Χόκμαρκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για την παρουσίασή της. Ένα πράγμα ήθελα να θέσω, για ένα ερώτημα για τα επόμενα βήματα. Παρουσιάστε την πρόταση για τον κανονισμό, για, το, για την περιεγωγή. Έχουμε και την ε, πολιτική για το νεοφάσμα και πρέπει βεβαίω να σκεφτούμε τι γίνεται παραπέρα για να μην χάσουμε και την, ε, το ορόσημο αυτό. Έχοντα υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με το, με το πιο σύγχρονο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας, μάλλον είναι παράδοξο ότι σε αυτό το τμήμα της οικονομίας έχουμε 27 μεμονωμένες επιμέρους αγορές, που αυτό αποτελεί πρόβλημα μένα, αλλά αποτελεί και ρίζα προβλήματος άλλων, και ρίζα άλλων προβλημάτων, συγγνώμη. Υπάρχουν λοιπόν και τρόποι ε, να λυθούν, ε, να, για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, απλή στον ορισμό τους, καθόλου απλή στην εφαρμογή τους. Ας πούμε το θέμα της αδειοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή αν μπορέσουμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο φάσμα για την ε, κυκλοφορία των δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα. Και αυτό θα αποτελέσει μια θετική εξέλιξη. Υπάρχουν λοιπόν πολλές, πολλοί τρόποι για να λυθεί αυτός ο κατακαιρματισμός. Οπότε το ερώτημά μου είναι πώς θα σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι 27 διαφορετικές αγορές. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ο πύρινας της δουλειάς σας τελικά. Ευχαριστώ. Εντάξει, ε, μια μισή ερώτηση από τον κύριο Χόκμαρκ. Λοιπόν, να δώσουμε τώρα το λόγο στην Επίτροπο για να προσπαθήσει να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας ξεκινήσω με εκφράζοντας πόσο ευτυχής είμαι για τα σχόλιά σας και για τη στήριξη της Επιτροπής Ήτρε για το θέμα της ε, περιαγωγής και το θέμα του φορέα ενισά του οργανισμού. Αυτό που θέλω να τονίσω και έτσι ε, απευθύνομαι και στον κύριο Χαλκμαρκ, ε, πράγματι ε, είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση βραχυπρόθεσμα. Ε, ο δρόμος έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Να επανέλθω λίγο όμως σε κάτι που είπα στην αρχή. Υπάρχει ελπίδα και κάτι παραπάνω από ελπίδα. Υπάρχει η ευκαιρία να δείξουμε και στον πολίτη, γιατί η πολίτης έχει αρχίσει να χάνει την κατεύθυνση ε, αμφιβάλλει αν υπάρχει ελπίδα. Εμείς μπορούμε να το αποδείξουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Αυτό που διακυβεύεται είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μειονέκτημα στον χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά αυτό μπορεί να μεταμορφωθεί και σε πλεονέκτημα. Με αυτό το οριζόντιο χαρτοφυλάκιο, με τη βοήθεια τη δική σας, με τη βοήθεια των συναδέλφων μας, πρέπει λοιπόν να το σμπρώξουμε. Γιατί επειδή είναι οριζόντιο, συνδέεται με πάρα πολλούς τομείς και πράγματι μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που απαιτείται και που είναι και, και που υπάρχει κιόλας. Ε, ε ανταγωνιστικότητα. Πολλές φορές μας κατηγορούν ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή νησίδα ε, και πολλές φορές όμως στις συζητήσεις μας βλέπουμε με τους συνομιλητές μας ότι και εκείνοι θεωρούν πως υπάρχουν ευκαιρίες και αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, να υποφεληθούμε. Το να ονειρευόμαστε μια ενιαία αγορά, μια ψηφιακή ενιαία αγορά, ε, είναι μια πραγματικότητα ακόμα και αν οι πολιτικοί και οι πολιτικοί θεσμοί δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να υλοποιήσουν την κατάσταση. Στην καθημερινότητά μας ήδη έχουμε μια ψηφιακή ενιαία αγορά, μια ε, ασύνοριακή αγορά, μια αγορά χωρίς σύνορα. Τούτου λεχθέντος, ε, επειδή μιλούμε για λιγότερους φραγμούς και λιγότερα σύνορα, ε, στις προτάσεις που παρουσίασα και χάρη σε εσά που με κρατάτε σε εγρήγορση και μου δίνετε ευκαιρίες και πρέπει να πω ότι ε, πολλές φορές θέλω να το πω αλλά δεν μου δίνετε την ευκαιρία. και δεν τολμώ να πω ότι υπάρχουν ευκαιρίες στην πραγματικότητα. Η κυρία Ντεκαστήγιο μίλησε για το υπολογιστικό σύννεφο, το cloud computing, για να είμαι απολύτως ανοιχτή μαζί σας. Για να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να το ολοκληρώσω μέχρι το 2012. Το υπολογιστικό σύννεφο διακυβεύεται παγκοσμίω και αν πρόκειται να παίξουμε όχι απλώς ένα ρόλο ως Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Αναμφίβολα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ψηφιακό μας μέλλον. Εξίσου σημαντικό είναι και για τον κλάδο, για τη βιομηχανία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τα άτομα. Ναι, αν επιτύχουμε να δημιουργήσουμε το δικό μας κλάδο, το δικό μας σύννεφο, το υπολογιστικό, θα είναι πολύ καλό. Και υπάρχουν ήδη μερικοί παίκτες που θα, θα ήταν ίσως ενδιαφέροντες εταίροι. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ε, ξέρετε τι είναι το υπολογιστικό σύννεφο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των φραγμών, μεταξύ των οποίων η ανεπαρκείς ή μη επαρκώς σαφής κανονισμοί για τα δεδομένα, την προστασία τους, την ασφάλειά τους, την ε, ευθύνη περί των σχετικών παραβιάσεων των σχετικών αρμοδιοτήτων δεν μας παίρνει να κάνουμε λάθος στον τομέα αυτό γιατί διαφορετικά θα ήταν σαν να ε, είμαστε σε τρίπια βάρκα. Πρέπει και πραγματικά εργαζόμαστε σκληρά ε, για να το επιτύχουμε. Ε, εργαζόμαστε με βάση όλων των απαντήσεων, άνω των 500 απαντήσεων, μετά, τον, μετά την δημοσίευση ενός σχεδίου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τον περασμένο Γενάρη. Ε, το οποίο το ανοίξαμε μαζί με άλλες διαδικασίες διαβούλευσης το 2011. Ε, ετοιμάζουμε την στρατηγική μας, ετοιμάζουμε το έγγραφο αυτό, το οποίο και θα αναλύει και θα προτείνει. Και υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να το έχω έτοιμο, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μην με κατηγορήσετε όμως αν βγει λίγο αργότερα. Για μένα το 2012 είναι πολύ σημαντικό να μπορέσω να το παρουσιάσω με ασφαλή τρόπο, για να το θέσω έτσι. Για την ψηφιακή ενιαία αγορά τώρα, η κυρία Χόλ, η κυρία Βέλιεν το έθιξαν. Πράγματι, πρέπει ε, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι σαφέστατο. Ναι, μιλήσατε και για τους επιχειρηματίες της Ευρώπης και για ανάπτυξη, γιατί πραγματικά έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Μέχρι στιγμής, για να το θέσω διπλωματικά, δεν έχει χρησιμοποιηθεί 100% αλλά πραγματικά αυτοί θα πρέπει να παίξουν το παιχνίδι και ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Πρέπει λοιπόν πραγματικά οι κανόνες μας να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή. Οι κανόνες για την επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων στοιχείων, ε, η πνευματική ιδιοκτησία, ε, η ηλεκτρονική ταυτότητα, η ηλεκτρονική υπογραφή. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Πρέπει να επιταχύνουμε μαζί με τους συναδέλφους μου. Χρειάζεται πραγματικά επιγόντως και ελπίζω ειλικρινώς να μπορέσω να βασιστώ και στη δική σας στήριξη και έτσι να μπορέσουμε πραγματικά να προχωρήσουμε στο ψηφιακό μας δρόμο ε, και να προχωρήσουμε τις προτεραιότητές μας. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, υπογραφή, πιστοποίηση, πραγματικά. Θα είναι μια ευρωπαϊκή στρατηγική όπως και με το υπολογιστικό σύννεφο. Και πάλι το 2012. Τώρα, το, οι δορυφορικές ε, οι κινητές υπηρεσίες. Στην ε, απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπάρχει πραγματικά απόφαση για να δημιουργηθεί ενιαία αγορά για το τομέα αυτό. Δεν, περαιτέρω συμφωνία από αυτό δεν επετεύχθη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμπορική ανάπτυξη των δορυφορικών κινητών υπηρεσιών όπως προβλεπόταν από το σχετική απόφαση και αυτό παρά την αύξηση της ζήτησης ε, για φάσμα. Αν υπάρχει αύξηση λοιπόν ζήτησης ραδιοσυχνοτήτων και φάσματος, πρέπει να <clears throat> το δώσουμε. Μας πιέζει ο χρόνος και δεν μπορώ να επεκταθώ. Τώρα, τον Οκτώβριο, η Επιτροπή υιοθέτησε μια απόφαση που της επιτρέπει να συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να ε, εφαρμόσουν στην πράξη τις ε, ε, υπηρεσίες αυτές. Διαφορετικά οι ραδιοσυχνότητες θα δοθούν για άλλο σκοπό. Και εσείς, ο κύριε Πρόεδρο και η κυρία Μέρκες και η κυρία Βάλιαντ μιλήσαν για την περιαγωγή. αναφέρεται, κύριος Τσίσεστερ το ανέφερε νομίζω. Ε, ε, το θέμα είναι πάντα να υπάρχει ανταγωνισμός ή ότι δεν υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός. Την τελευταία φορά ε, διαπιστώθηκε ότι εποφελήθηκαν οι καταναλωτές, αλλά είδαμε ότι το μέρος του, του ανταγωνισμού παραμελήθηκε ίσως και πρέπει να το προσέξουμε. Να διευκολύνουμε την είσοδο των νέων παικτών, να αυξήσουμε την επιλογή των, των καταναλωτών. Με συγχωρείτε. Ε, πραγματικά καλό θα ήταν ε, ο υποψήφιος πελάτης να έχει πραγματικά τις επιλογές που αναφέρεται, αλλά ας ξεκινήσουμε και θα δούμε που θα πάμε και νομίζω ότι η πρόταση αυτή αποτελεί ένα πρώτο μεγάλο ε, βήμα. Τα ανώτατα όρια των τιμών τα χρειαζόμαστε προς το παρόν, θα ήταν ρηψοκίνδυνο να τα εγκαταλείψουμε. Ε, ε, πού βρισκόμαστε τώρα με βάση με την στενή συνεργασία και θέλω να το αναφέρω και πάλι ε, είμαστε σύμμαχοι και θέλω να προχωρήσουμε έχουμε υποσχεθεί ε, να επιταχύνουμε την καινοτομία ε, για να ανταποκριθούμε και στην αλλαγή της δημογραφικής κατάστασης, τη γύρανση του πληθυσμού. Το λαμβάνουμε υπόψη. Και <clears throat> θα ελπίζω για όλους μας ε, να έχουμε χρόνια υγιή και περισσότερα μπροστά μας. Υπάρχει συνέργεια μεταξύ ε, των εμπλεκόμενων πλευρών και πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς. Στην περίπτωση αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία στην πολιτική μου ζωή που οι Υπουργοί Οικονομικών είναι φίλοι μου. Μακροπρόθεσμα πραγματικά θα αναγνωριστεί αυτό, ότι με την ενισχυμένη συνεργασία και με την εισαγωγή των ψηφιακών ευκαιριών θα πληρώνουν όλοι φθηνότερους λογαριασμούς, για να το θέσω έτσι απλά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη στήριξή σας. Η Ενισά. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις όλων. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για τον εξυγχρονισμό και την ενίσχυση της ΕΝΙΣΑ. Αυτό που θέλω να αναφέρω, κύριε Πρόεδρο, είναι ότι όταν ο οργανισμός αυτός ξεκίνησε, ήταν λίγο διαφορετική η εποχή. Όπως και να έχει, δεν γνωρίζαμε τότε αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Την εποχή εκείνη δεν ήμασταν ικανοί να ονειρευτούμε, αν θέλετε, αυτά που γίνονται σήμερα. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε τι πρέπει να εγκαταλείψουμε και τι πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο και τι ζητάμε από τον οργανισμό αυτό να κάνει. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο ε, για να καταστεί, πιο ασφαλές το ψηφιακό περιβάλλον στην Ευρώπη για τους πολίτες, τους πελάτες, ε, τις εταιρείες. Ε, μιλώ ο κάθε Ευρωπαίος να γίνει ψηφιακός. Ε, μου λένε να γίνουμε όλοι ψηφιακοί, αλλά με την ασφάλεια τι γίνεται. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση. Αλλά δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν μια απειλή. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε σαν ευχαρίστηση, σαν ευκαιρία. Πολλά λοιπόν μένουν για να κάνει ο οργανισμός αυτός. Και ορθά επεσήμανε ο πρόεδρος ότι πώς μπορείς να προσελκύσεις τους καλύτερους ανθρώπους που τους χρειάζεσαι. Αυτό φυσικά και με μεγάλη προσοχή το αναφέρω. Πριν αρχίσετε να γελάτε, χθες ε, μιλούσαμε νέους επιχειρηματίες ε, μέλη διοικητικών συμβουλίων και ανώτατα διευθυντικά στελέχη και με παρουσίασαν και είπαν ότι όταν για πρώτη φορά έγινα βουλευτής ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, αυτοί δεν είχαν καν γεννηθεί και γελούσαν όλοι. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν είναι μόνο η ενισά. Ε, όλος ο κόσμος χρειάζεται ένα περιβάλλον ασφαλές, όπου να υπάρχει πρόσβαση ε, όχι μόνο για, τους, για τον κάθε άτομο μεμονωμένα, αλλά και για την οικογένειά του. <clears throat> Όπως και να είναι. Πρέπει να ξέρουμε ότι ε, μιλάμε για τα πρώτα βήματα. Μόλις τώρα στείλουμε την ομάδα στην Αθήνα, είναι ένα πρώτο βήμα και με την ε, ομάδα ε, κινητής ε, βοήθειας θα προχωρήσουμε και ελπίζω πραγματικά το επιχειρησιακό κέντρο να μείνει στην Αθήνα. Δεν θέλω να φύγουμε από την Ελλάδα. Καθόλου. Αλλά να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό μοντέλο. Να τους βάλουμε κάπου από όπου να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Δεν μου μιλάει χωρίς να λέει κάτι συνέχεια. Δεν μπορώ άλλο να εφεύρω νοήματα. Για, ε, για, την... για την ουδετερότητα του δικτύου. Ε, πραγματικά είμαι Αφοσιωμένη στη διατήρηση του ανοιχτού χαρακτήρα του διαδικτύου. Πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ε, σε ανταγωνιστικές αγορές. Πάντοτε το επαναλαμβάνουμε. Αν υπάρχει ανταγωνιστική αγορά, τα πράγματα λειτουργούν για τον καταναλωτή, για το μέλλον, για την έρευνα, για την καινοτομία, για όλα. Αλλά για να λειτουργήσει σωστά ο ανταγωνισμός, οι πελάτες θα πρέπει να είναι ικανοί και σε θέση να, κάνουν, να λαμβάνουν αποφάσεις με τα λόγου γνώσης. Και εδώ η λογοδοσία και η διαφάνεια παίζουν ρόλο. Θα πρέπει να μπορούν να αλλάξουν πάραχο υπηρεσιών άνετα και γρήγορα και εύκολα. Εάν ε, προσφέρεται η δυνατότητα να αλλάξει, αλλά είναι γραφειοκρατική και παίρνει ένα σωρό χρόνο, δεν έχει νόημα. Επίση, πρέπει οι ρυθμιστικέ αρχέ να έχουν μια εργαλειοθήκη, κάποια μέσα στη φαρέτρα του. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να, το, να παρατηρούμε την κατάσταση και αν τα καινούργια μέσα δεν είναι επαρκή να λάβουμε και άλλα μέτρα. Α Ας είμαστε λοιπόν ανοιχτοί. Ποια είναι η άποψή σας για την Ολλανδική πρόταση. Ο κύριος Χράουτε έκανε την ερώτηση. Εγράψαμε στις Ολλανδικές Αρχές και σας ενημέρωσα και νωρίτερα και ζητήσαμε περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο νόμου τους. Αυτό είναι νομίζω επαγγελματικό. Ε, μπορεί κανείς να το κάνει. Ε, Σημερίζομαι τις ανησυχίες των καταναλωτών, των βουλευτών επίσης, για τον αποκλεισμό διαδικτυακών υπηρεσιών. Πρέπει να δράσουμε συντονισμένα σε όλη την Ευρώπη. Και γι' αυτό ζητώ από τον Μπέρεκ ε, το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο να συστήσουν ένα φορέα που να είναι ανεξάρτητος και να μπορεί να παρέχει συμβουλές και ζητώ λεπτομέρειες και παρακαλώ πάντοτε θέλω να είμαι σε επαφή με την πραγματική ζωή και περιμένω μέχρι να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί διαφορετικά αν οικοτολογώ και λέω ναι νομίζω ότι ε, τότε δεν είμαι δίκαιη απέναντι στον Μπέρεκ και δεν είμαι και επαγγελματία. Ασφάλεια. Κυρία Μαντερέλ, αναμφίβολα η στρατηγική ασφάλεια του Ευρωπαϊκού Δαδικτύου ε, και συνδέεται στενά και με τον ΕΝΙΣΑ ε, πρόκειται να στηθεί μέχρι το 2015 και ελπίζω μέχρι τότε να έχουμε σωστή άμυνα. Μέχρι τότε θα δεχτούμε κυβερνοεπιθήσεις, κυβερνοεπιθέσεις. Πρόσφατα ε, πάλι είχαμε κάποιες εμπειρίες, οπότε ξέρουμε τι διακυβεύεται και πρέπει πραγματικά να έχουμε ε, ε, ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών ασφάλειας του κυβερνοχώρου, να έχουμε ε, σχέδια για έκτακτες παραβιάσεις, οργανωμένα δίκτυα, οργάνωση ασκήσεων και επίσης να είμαστε πάρα πολύ ενεργοί στην συνεργασία μας με διεθνείς παίκτες και εταίρους. Στον τομέα αυτό είναι σαφές ότι δεν σταματάει η απειλή στα σύνορα. Επομένως χρειαζόμαστε στενή συνεργασία και με τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και με άλλες πλευρές. Σχεδόν τελείωσα. Α, το Connecting Europe Facility, το μέσο για σύνδεση της Ευρώπης. Με ρωτήσατε πώς Αναμένω, μήπως περιμένω να δω προς τα που θα φυσήξει ο, άνεμος. Ε, ε, είμαι σοβαρή όταν μιλώ για 7 δισεκατομμύρια από τα 9,2 δισεκατομμύρια για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και για τις υποδομές. Και όλη αυτή η μόχλευση που ανέφερα είναι ευσεβής πόθη ή σοβαρόλογο. Σοβαρόλογο, σοβαρόλογο απόλυτα Έχουμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουμε συζητήσει μαζί τους και με άλλους. Δεν μιλούμε μόνο για κάποιον επενδυτή, αλλά και άλλες πλευρές. Πρόκειται για σοβαρή πρόταση. Με τη μόχλευση μπορείς όντων να φτάσεις μεταξύ των 60 και των 100 ε, δισεκατομμυρίων. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε και στα 100 δισεκατομμύρια. Να πάμε βέβαια, οι άλλοι με προειδοποιούν, μου λένε πρόσεχε τα λόγια σου, μην... ας πάμε στη μέση, ας το σπάσουμε στη μέση. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν πολίτες, τα δικαιώματά τους από την ελευθερία έκφρασης μέχρι την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ελάχιστη εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών. Ξέρουμε ότι τα δικαιώματα αυτά είναι σκόρπια και κατατετμημένα στα διάφορα δίκαια και δεν είναι πάντοτε εύληπτα και αυτό για τον καταναλωτή, τουλάχιστον έτσι έχουμε μάθει, ε, καθιστούν τον καταναλωτή ανίκανο να εκμεταλλευτεί πλήρως την ψηφιακή αγορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, και ένα ψηφιακό δικαίωμα υποβολής παραγών, παραπόνων. Τώρα για την ε, ε, συμμετοχή των γυναικών ε, γνωρίζω πολύ καλά ότι χρειαζόμαστε τις γυναίκες στην τεχνολογία. Αν σας δώσω τους αριθμούς των προγνώσεων 7-8 χρόνια από τώρα για τον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, πραγματικά χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους και και κανένας δεν μπορεί να πει ότι όχι, μόνο ένα κομμάτι του ανθρωπίνου είδους θα συμμετέχει. Τι διακυβεύεται. Και αυτό πραγματικά είναι συναρπαστική πρόκληση. Σε οκτώ χρόνια από τώρα, ή σε 10 χρόνια από τώρα. Αν θέλεις αποτελέσματα σε 8 με 10 χρόνια από τώρα, πρέπει να ξεκινήσεις από τώρα. Είναι μια διαφορετική νοοτροπία. Πρέπει να ξεκινήσουμε με την νεότερη γενιά γυναικών. Δεν θέλω να μιλήσω για τους αριθμούς. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Χρειαζόμαστε εντυπωσιακό αριθμό και από τις επιχειρήσεις ε, που μας ενημερώνουν. Δεν μιλούν μόνο για μηχανικούς ε, πληροφορικής, αλλά ε, όλες οι ειδικότητε πολλές ευκαιρίες λοιπόν. Γι' αυτό πραγματικά με έχει συνεπάρει αυτός ο τομέας και... και... Ε, Θέλω, έρχο, είμαι σε επαφή και με, τις, ε, με τους οργανισμούς απασχόλησης εργατικού δυναμικού. Εάν μπορεί κανείς να εστιάσει την προσοχή του σε αυτήν την ομάδα και στην νεότερη ομάδα ακόμη αν έχουμε τόσους πολλούς άνεργους νέους, μπορείτε να φανταστείτε ε, τι μπορούν να ελπίζουν και να σκέφτονται οι ακόμη νεότεροι από τους νέους ανέργους. Πρέπει λοιπόν να την εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και νομίζω ότι η τεχνολογία αυτή για τις γυναίκες είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να, στα οποία, πάνω στο οποίο πρέπει να ενσκύψουν πολλές πλευρές, όχι μόνο η Επίτροπος την, για το ψηφιακό θεματολόγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούμε να πούμε ότι είναι ο ψηφιακός πρωταθλητής γιατί το διασυνδέει με την ε, εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση που δείχνει πόσο ελκυστικοί μπορούμε να γίνουμε ε, σε αυτές τις θέσεις εργασίας. Μπορεί να ζητήσω και από τον Πρόεδρο να γράψει μια επιστολή σε όλα τα κράτη-μέλη, στους Πρωθυπουργούς και τους Προέδρους και να τους ζητήσει να, διορίσουν και αυτοί έναν τέτοιο πρωταθλητού όπως η Μάρθα αν θέλετε. Αν μπορείτε να κάνετε τον πρωθυπουργό σας ή τον πρόεδρό σας να πανηγυρίσει αυτή την ιδέα μιας ε, γυναικείας μορφής πρωταθλήτριας στο ψηφιακό τομέα θα ήταν πολύ καλό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για τις πληροφορίες σας, για τις απαντήσεις σας στα ερωτήματά μας. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες φαντάζομαι θα είμαστε σε στενή επαφή γιατί ακόμα υπάρχουν πολλά θέματα εκκρεμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.